Okay, colleagues, we're going to begin our afternoon session. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον ε, των σχέσεων ΑΣΕΠΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με γνωρίζετε, είμαι πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα προεδρεύσω στην έναρξη και μετά θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο του Φρανκ Έγκελ που είναι εδώ στα αριστερά μου και εγώ θα τα αφήσω στο κοινό για να παρακολουθήσω τι παρουσιάσει. Για την Επιτροπή μας ε, το θέμα αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα Γι' αυτό ακριβώς ε, και είναι μεγάλη χαρά να έχουμε τόσο εγνωσμένου κύριους ε, προσκεκλημένους εδώ. Έχουμε καταρχάς ε, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ, το Κεν Ντούνς. Έχουμε τον μου Γκομετζούλου, πρέσβη της Σουαζιλάνδης, η πρόεδρο της Επιτροπής Πρέσβεων των Χωρών ΑΚΕ. Βιβανού Νασούνου, ε, βοηθός ε, γενικός γραμματέας ε, των, ε, της ομάδας χωρών ΑΚΕ. Θα σας κάνω μια εισαγωγή. Έχουμε αρκετούς ομιλητές. Θα τους παρουσιάσει βέβαια ο ε, συντονιστής του κάθε πάνελ, ε, δεν χρειάζεται να σας τους συστήσω εγώ. Εγώ απλώς ε, θα ε, κάνω μια αρχική παρουσίαση εκ μέρους Επιτροπής. Είναι πολύ καλή στιγμή η σημερινή συγκυρία για να γίνει αυτή η συνεδρίαση, γιατί όπως γνωρίζετε το σχέδιο εντολής για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπεται να εγκριθεί φέτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και από τους Υπουργούς ε, στο Συμβούλιο και οι επίσημες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Ως Επιτροπή Ανάπτυξης συμφωνήσαμε να καταθέσουμε μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους συναδέλφους η αγγλική εκδοχή βρίσκεται στους φακέλους σας και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή ΔΕΒΕ του Απριλίου. Προθεσμία για τις τροπολογίες ε, σημειώστε παρακαλώ. Παρασκευή 6 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Πριν δώσω το λόγο στους συντονιστές ε, των δύο πάνελ, θα ακούσουμε μία ε, γενική παρουσίαση από τον καθηγητή Λούντγκερ Κρούνχαρντ, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου για τις ε, ε, ε, ε Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ε, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες. Καθηγητή Κρούνχαρντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη. Ε, πρέσβης ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εντολή για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ομάδα χωρών ε, ΑΚΕ που δημοσιεύθηκε το 2017 είναι πιο φιλόδοξη από ό,τι περίμεναν πολλοί. Είναι πολύ καλύτερη και σε περιεχόμενο και σε γλώσσα, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης βεβαίως και πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε ε, την πολιτική φιλοδοξία, το στρατηγικό μας σχεδιασμό, αναφέρεται σε κοινέ αξίες και όσο καλά είναι αυτά, ε, τέτοιες ε, απαριθμίσεις στοιχείων είναι απλώς ένας κατάλογος επιθυμιών, ένα ευχολόγιο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, να είμαστε ειλικρινεί ε, για τα εμπόδια, λέει πολύ συχνά η πρόταση και τα προσκόμματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά υπάρχει και ε, ένας κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει μονίμως και φαίνεται σε όλο το κείμενο ότι μπορεί να επαναλάβουμε τα ίδια πράγματα. Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις βασικές πτυχές, οι οποίες ε, πρέπει να αναλυθούν περισσότερο στι ε, μελλοντικέ συζητήσει ε, που θα κάνετε και στην Επιτροπή ανάπτυξη. Καταρχά, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να υπάρχει μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Ο στόχο θα είναι, όπω λέει η πρόταση και σα παραθέτω, μια νέα συμφωνία η οποία θα αποτελείται από τρει ε, περιφερειακέ συμφωνίε που θα βασίζονται σε κοινά θεμέλια. Προτάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα ε, για ένα περιφερειακό σύμφωνο με την Αφρική, για την Καραϊβική ε, και για τις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ συγκεκριμένε σε κάποιες περιπτώσεις. Η πρόταση δεν ε, ε, υπερβάλλει διευρύνοντας ε, περαιτέρω στη Λατινική Αμερική και στη Νότια Αφρική, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δύο περιοχές. Για παράδειγμα, ε, κάποιες επιπέρων περιφερειακών ε, συμφώνων που θα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των διαφορών χωρών, των ομάδων χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τα θεμέλια όμως είναι ως προς την ουσία και τη σημασία τους λίγο αδύναμα. Ε, οι αρχηγοί κρατών και ε, κυβερνήσεων κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν να συμβάλλουν σε σημαντική καινοτομία στη συνολική διακυβέρνηση. Αν γίνουν καλά όλα αυτά και ίσως είναι καλύτερα από όσα αναφέρονται μέχρι τώρα, αυτά τα κοινά θεμέλια θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τη βάση για ουσιαστική καινοτομία στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά. Ε, προτείνω μία ε, συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χωρών και νομίζω ότι η Επιτροπή σας θα προτείνει κάτι ακόμα πιο ισχυρό με στόχο και πάλι να αναφερθούμε στη διαδικασία, να αναφέρουμε τις σχετικές πόλεις για να μπορέσουμε να δώσουμε και την κατάλληλη πολιτική ε, διάσταση και να έχει και το κατάλληλο εμπορικό όνομα εντό αγωγικών αν θέλετε. Ο στόχος της νέας ε, συνθήκης, ε, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι να υπάρχει μια πολιτική εταιρική σχέση για να δημιουργήσουμε μια ειρηνική, σταθερή, καλή διακυβέρνηση και να έχουμε ε, πόλεις και κοινωνίες που ευημερούν. αληθεύει μεν αυτό, αλλά κοιτάει μόνο την πλευρά της εταιρική σχέσης ε, των χωρών και. Δεν ξέρω αν απευθύνεται και σε εμά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ακούμαστε ε, ευημερία και ανθεκτικότητα και κοινωνίες. Ε, πρέπει να υπάρχει στήριξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν οι στόχοι είναι και προς τον συμφέρον των περιοχών ε, των χωρών ΑΚΕ, αλλά και προς τον συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών τους. Η γεωπολιτική σημασία μιας ανανεωμένης εταιρικής σχέσης είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίως αν ε, λάβουμε υπόψη τα 27 σύντομα κράτη-μέλη, ε, και τις 29 χώρες εάν ενταχθεί και η Κούβα, χώρες ΑΚΕ, και θα έχουμε δηλαδή ε, ε, πολύ μεγάλο αριθμό χωρών στα Ηνωμένα Έθνη και έτσι θα είναι στρατηγική σημασία στα Ηνωμένα Έθνη και στο σύστημα αυτό για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το σκοπό μας. Μήπως θα ήταν λογικό, για παράδειγμα, να υπάρχει ε, ένα τμήμα συντονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και στην, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ερωτηματικό εδώ. Θα πρέπει να δεχτούν την επιθυμία των χωρών ΑΚΕΝ να συμμετέχουν με άλλους εταίρους παγκοσμίω, ανεξάρτητα από τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, υποστηρίζοντας αυτό το ένομα συμφέρον των περιοφεριών ε, των χωρών ΑΚΕ και των ομάδων που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κατά την ταπεινό μου γνώμη να ε, ζητήσει ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητών ε, για τις ε, κυρίαρχες περιφερειακές ομάδες της περιοχές των χωρών ΑΚΕ, όπως είναι και το αναβαθμισμένο καθεστώς παρατηρητή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω σταθερότητα. Αυτό χρειάζεται να υπάρχουν παράγοντε που θα μπορούν να ε, αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να δημιουργήσουν και νέους κανόνες. Η νέα συνθήκη θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα αυτής της φύσεως, ενώ οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ Εθνών περιλαμβάνουν αρκετέ αντιφάσει, ε, στόχου που δεν συνάδουν μεταξύ του και έχουν μηχανισμού που δεν ε, ταιριάζουν απολύτω, θα μπορούσε η νέα συνθήκη να είναι μια ισχυρή, πολυμερές και ε, ίσως και η μόνη σημαντική προσπάθεια για εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας ε, μεταξύ των χωρών. Αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ ε, στην παγκόσμια τάξη ε, και φυσικά ίσως θα μπορούσε να είναι και μια λύση για να διατηρήσουμε και τη συνοχή των χωρών ΑΚΕ. Να προωθήσουμε από κοινού ε, μια ε, σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση ίσως ε, θα ήταν κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού. Τρίτον, το Brexit. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ασχολείται πουθενά την, με την πιθανή αποδόμηση που μπορεί να υπάρξει λόγω του Brexit και το πώς θα επηρεάσει την ομάδα χωρών και τι συνέπειες και τι αντίκτυπο θα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο φαίνεται να πλανάται και δεν είναι και τόσο διπλωματικό να το πω η Αφρική θα προτιμήσει περισσότερο τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ή με τη σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Και επίσης, οι μικρότερες και πιο απομακρυσμένες περιοχές είναι ίσως αυτές οι οποίες θα πληγούν περισσότερο. Το πρώτο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης που έλαβα μετά από το δημοψήφισμα ε, ήταν από τα νησιά Φίτζι. Τι θα γίνει με τη σταθερότητα στο Φίτζι, ε, αν υπάρχουν δασμοί και ποσοστώσεις για τις μελλοντικέ εξαγωγές Ζάχαρη μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και πώ οι χώρες θα οργανώσουν το μέλλον τους ε, ε, όταν είναι και χώρες που ανήκουν και στην κοινοπολιτεία. Ε, έχει πεθάνει αυτή η ιστορία, ενώ οι χώρες της κοινοπολιτείας ε, θα έχουν περισσότερο ημόχλευση εάν δεν κυρώσουν αυτό που έχουν ήδη ε, υπογράψει γιατί δεν το πιστεύουν ή γιατί φοβούνται. Και τι θα μπορέσει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους διστακτικούς εταίρους μετά τον Brexit. Και κάτι που ξεχνάμε συχνά, τι θα γίνει με τις υπερπόντιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδάφη μετά το Brexit. 12 από αυτές θα αποχωρήσουν από την Ένωση όταν θα γίνει το Brexit. Οι ε, υπερπόντιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται περισσότερο στην Ανταρκτική, ε, τα νησιά Φόκλαντ που ανησυχούν για τη μελλοντική πρόσβαση αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης η πρόσβαση στην Ανταρκτική που είναι πάρα πολύ σημαντική και το γεγονός ότι πρωτοπορεί σε θέματα κλίματος και σε γεωπολιτική. Ε, θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να ασχοληθεί και με τα θέματα αυτά σε πλαίσια ε, συζήτησης χωρών Και η πιο μεγάλη υπερπόντια περιοχή βρίσκεται στην Καραϊβική, ε, που έχουμε εκεί πολύ σημαντικές πτυχές για τη συνοχή της Κάρικο. Ε, αν ε, θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος μάλλον, υπάρχουν περιοχές στην Τζαμάικα για παράδειγμα, που φοβούνται ότι θα χάσουν τις δυνατότητες που έχουν και σκέφτονται να φύγουν και από την Caricom και ότι μπορεί να υπάρχουν συνέπειες στο εμπόριο λόγω του Brexit, ως άμεση συνέπεια. Καμία άλλη περιοχή και δεν περιλαμβάνει τόσες ε, υπερπόντιες ε, περιοχές και εδάφη και φυσικά οι χώρες ε, της Καραϊβικής κυρίως θα πληγούν λόγω του Brexit. Μπορεί να υπάρξουν και νέες... ε, ομάδες χωρών ε, στην όλη έννοια της ΑΚΕ και το θέμα της αμοιβαιότητας. Για παράδειγμα, χρηματοδότηση κοινή έρευνας ε, με χώρες της κοινοπολιτείας και για βρετανικές ε, υπερπόντιες περιοχές και δάφη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα νομίζω ότι οι συνέπειες του Brexit για αυτές τις υπερπόντιες περιοχές και δάφη, γι' αυτό και το θίγω, ε, είναι το βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και θα πρέπει ο γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ακόμα πιο λογικός. Και αυτό έρχεται να προσθεθεί και στα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι έτοιμα και ενωμένα για να ε, ε κάνουν επιτέλους έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τα ερωτήματα του Brexit απαιτούν μια πιο συνεκτική, πιο ενωμένη Ευρώπη. Και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνο να ασχοληθούμε με πολλά θέματα και πολλέ πτυχέ. Πολλά από αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε δε. Αλλά είναι και ζωτική σημασία ε, να καθορίσουμε βασικέ προτεραιότητε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο τέλο τη παρουσίασή μου θα σα τα παρουσιάσω επιγραμματικά. Αναπτυξιακή βοήθεια, η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους ΑΚΕ και την τελική ε, δημιουργία αυτής της σχέσης, η πρόκληση είναι να προσθέσουμε νέα αξία και να προσδώσουμε σημασία στην ίδια την έννοια της ανάπτυξης όλες οι χώρες της Γης και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ είναι αναπτυσσόμενες χώρες και η βοήθεια κατά την άποψή μου είναι παγκόσμια συμβολή στην ευημερία αλλά όχι ο κινητήριος μοχλός της ευημερίας. Και οπουδήποτε και να προχωρήσουμε, ε, δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε πλήρως ε, και πώς εφαρμόζουμε σε κάθε τομέα στους μηχανισμούς ρύθμισης και διακυβέρνησης. Αυτό αφορά πολιτικές κατά των μονοπωλίων, ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μην υπάρχει υπερβολική χρήση δημοσίων ε, ενισχύσεων κλπ. Και πρέπει φυσικά να δούμε και τι γίνεται με το περίπλοκο θέμα των δικαιωμάτων επί της γης και πρέπει να δούμε και τα επενδυτικά σχέδια. Δεύτερο, εμπόριο. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία που ελπίζω ε, να υπάρξει μια νέα συμφωνία στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρουσιάσει πιστικά επιχειρήματα για να βοηθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις και γιατί η προστασία των επενδύσεων και του εμπορίου είναι προς το συμφέρον όλων. Συμφωνώ με τον Γενικό Γραμματέα των χωρών ΑΚΕ, τον κύριο Γκόμες και παραθέτω στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις η ευρωπαϊκή πλευρά απέτυχε να διαρθρώσει και να κατανοήσει το εμπόριο ως ε, εργαλείο ανάπτυξης. Αυτό ισχύει κυρίως για μικρότερες και φτωχότερες ε, χώρες ΑΚΕ. Και όσον αφορά τη γεωπολιτική και το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε νέες μεγάλες αναδυόμενες αγορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ πρέπει να χρησιμοποιήσουν καλύτερα το τριμερές εμπόριο και τη συνεργασία με οποιαδήποτε τρίτη χώρα ενδιαφέρεται να συνεισφέρει στου στόχου που επισημαίνονται σε αυτή τη νέα πρόταση εταιρική σχέσης. Η ε, ροή εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και αυξήθηκε, διπλασιάστηκε από το 2000, είναι 5% των ευρωπαϊκών εξαγωγών και εισαγωγών και θα πρέπει να είναι κίνητρο αυτό για να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο δημιουργικοί χωρίς να υπάρχει και αίσθηση ε, ήτας, ε, ε, κυρίως όταν γίνονται συζητήσεις για την Κίνα. ο, τα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα σίγουρα θα αποτελέσουν κεντρικό κομβικό στοιχείο και δεν θα είναι συμπληρωματικό όπως προτείνεται στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σελίδα 42. Τρίτο και τελευταίο, πολιτική βούληση. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευρύ προτείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεράσει ε, τη παραδοσιακή νοοτροπία που έχει να δασκαλεύει τους, ε, τις χώρες ΑΚΕ και να τους επικρίνει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερο αμοιβέ διαδικασίες στον τομέα του πολιτικού διαλόγου, για παράδειγμα, και να ε, προσκαλέσει για παρακολούθηση εκλογών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκπροσώπηση των χωρών ΑΚΕ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε η εφαρμογή της μελλοντική συνθήκης ε, αναφέρεται για να αποφύγουμε ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων να μην δημιουργήσει μια ακόμα βιομηχανία ε, δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης που θα είναι αποδεσμευμένες και από την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ. Είναι απαραίτητος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σίγουρα. Η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι ευρύτερη στην πολιτική σφαίρα και θα πρέπει να είναι και πιο ε, εύρωστη και να έχουμε νέους τρόπους να προσεγγίσουμε την κοινωνία των πολιτών πέραν των παραδοσιακών ομάδων και ομάδων συμφερόντων. Σε επίπεδο κάθε περιφερειακού συμφώνου και σε συνολικά σε επίπεδο χωρών και. αλλά εδώ τίθεται το δίλημα του κινδύνου της επανάληψης και του κίνδυνου, κίνδυνου της έλλειψης ε, νομικά δεσμευτικά ε, μέσων για όλους. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσετε και στην Επιτροπή σας. Ε, φαντάζομαι ότι σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δομές όπως μια Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων Χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα φόρουμ μετανάστευσης, ε, ένα φόρουμ ε, ε, μελετών ασφαλείας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ήταν προνόμιο για μένα να σας απευθύνω το λόγο εδώ στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το 7,3% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι το 12% του παγκοσμίου ΑΕΠ και συμβάλλει το 35% του παγκοσμίου εμπορίου, η χώρα ΑΚΕ είναι το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού, 1,9% του ΑΕΠ κόσμου και συμβάλλουν 4,7% του παγκοσμίου εμπορίου. Σίγουρα λοιπόν αποτελούν διαφορετικές και ασύμετρες πραγματικότητες. Αλλά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ζωτική σημασία για τους επόμενους μήνες για να προωθήσει και να προωθήσει αυτή τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού ε, γι' αυτό που είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, μια πάρα πολύ σημαντική του παγκόσμιου σημαντικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια δοκιμή για το πώς μπορούμε να έχουμε ε, πολυεπίπεδη πολιτική σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προσφέρατε τροφή για σκέψη και για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση. Σήμερα το πρωί όλοι συμφωνήσαμε ότι θα συζητήσουμε για το Brexit σε βάθος. Θα μας άρεσε πολύ να έχουμε έναν αντίγραφο της ομιλίας σας για να επιλέξουμε κάποια θέματα. Ε, οι ερωτήσεις δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν όταν θα έχουν μιλήσει όλοι οι ομιλητές του πρώτου πάνελ, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Ως εκ τούτου ε, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έγγελ που θα προεδρέψει στο πρώτο πανέλ και εγώ θα πάω κάτω στα κάτω έντρανα για να παρακολουθήσω ως απλή βουλευτής. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ε, προχωράμε λοιπόν ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση διότι ίσως ε, ε, περιστούμε, ίσως αντιμετωπίσουμε πρόβλημα χρόνου και δεν θέλω να περικόψω το χρόνο των αγορητών που θα ακολουθήσουν. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο πάνελ, συνεχίζουμε με τις ομιλίες. Ξεκίνησε ο καθηγητής κύριος Κιούνχατ. Πρόκειται για την κατάσταση που θα ακολουθήσει μετά τις διαπραγματεύσεις ε, Κοτονού. Οκτώ λεπτά τα έχει ο καθένας από τους επόμενους ομιλητές. Αν έχει την καλοσύνη να τηρήσετε λιγάκι αυτό τον προβλεπόμενο χρόνο για να μην έχουμε στο τέλος ε, πίεση χρόνου και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Κιοντούν ε, που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ΤΕΦΚΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είχαμε τη συζήτηση να συζητήσουμε αρκετές φορές με την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, για την κατάσταση μετά το Κοτονού και χαίρομαι που ε, μπορούμε να δούμε λιγάκι το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Ευχαριστώ και τον κύριο Κούνχαρτ για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του. Είπατε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ καλύτερη από την αναμενόμενη. Δεν ξέρω αν το θέλετε, αλλά εγώ θα το εκλάβω ως φιλοφρόνηση. Συμφωνώ με την πρόταση. Ε, θέλω βέβαια να υπογραμμίσω ότι και ο, ο, ο Επίτροπος Μιμίτς ε, στις 25 Ιανουαρίου παρουσίασε την πρόταση Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Ανάπτυξης και καταλήξαμε ε, στο ότι ευθυγραμμίζονται οι απόψεις των Ευρωβουλευτών και της Επιτροπής. Σύντομα λοιπόν θα μιλήσω για το τι έχουμε προτείνει, γιατί το προτείναμε και επίση ε, και γιατί τα πάμε αρκετά καλά στο να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο, αυτό να το πετύχουμε το Μάιο ε, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η πεμπτουσία της πρότασής μας είναι, όπως γνωρίζετε, να δημιουργηθούν ισχυρά θεμέλια και πάνω σε αυτά τα θεμέλια που αφορούν το σύνολο των χωρών και πάνω σε αυτά να οικοδομήσουμε ουσιαστικά τρία σπίτια, τρεις ε, πυλώνες, ένας με την Καραβική, ένας πυλώνας με την Αφρική και ένας άλλος με τον Ειρηνικό. Πρόκειται λοιπόν για μια λύση που αντικατοπτρίζει τόσο τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες όσο και την δύναμη της σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ΑΚΕ. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι πολύ απλός. Ξεκινάμε με γεωπολιτική διάσταση. Η γεωπολιτική διάσταση σε έναν πολυπολικό κόσμο νομίζω θα ήταν παραφροσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρετηθεί από αυτήν την ε, μακροχρόνια στρατηγική και σημαντική σχέση που έχει με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό χωρών στον κόσμο. Ε, και με τις χώρες αυτές έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο. Επιπλέον, η Ευρώπη έχει εμπλακεί σε αυτό τον πολυπολικό κόσμο με αυτό που είχε πει ο στρατηγός Ντεγκόλ σε ελεύθερη μετάφραση ε, μια συγκεκριμένη ιδέα της ε, Γαλλίας, ε, να το πούμε μια συγκεκριμένη άποψη για το πώς ε, λειτουργεί ο κόσμος. Έχουμε μια τέτοια άποψη και δεν ε, συμπίπτει απαραίτητα με την άποψη των υπόλοιπων υπερδυνάμεων στον κόσμο. Ξεκινάμε από αυτή τη βάση για τις σχέσεις με τις χώρες και αυτό για μας ήταν καθοριστική σημασία. Βεβαίως έχουμε ένα ε, πολύ ε, καλό πλαίσιο ότι το θεματολόγιο του 2030 πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τη σχέση μας σε αυτό το νέο διεθνές θεματολόγιο. Ο κύριος καθηγητής έκανε αναφορά στα συμφέροντά μας. Πράγματι έχουμε δικά μας συμφέροντα και το ίδιο ισχύει και για τις χώρες ΑΚΕ. Νομίζω λοιπόν σε αυτό το νέο πλαίσιο μπορούμε να είμαστε περισσότερο σαφείς ε, για το ότι αυτή η νέα ρύθμιση προβλέπει τη σύγκληση των συμφερόντων. Έχουμε εντοπίσει προτεραιότητες οι οποίες με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν αυτονόητες αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αυτονόητες ε, δεν είναι και σωστές και επειδή είναι σωστές δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικές. Νομίζω ότι οι ομάδες που έχουμε εντοπίσει, ε, διαχείριση, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, ασφάλεια, ανάγκη να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, η ανάγκη να υπάρξουν επενδύσεις σε άτομα, στην ε, ανάπτυξη του ανθρώπινου στοιχείου, να αντιμετωπίσουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μετανάστευση και κινητικότητα. Να δούμε πώς μπορούμε να δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων ε, και τέλος ε, το πώς μπορούμε όλοι από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας που είναι η κλιματική αλλαγή, ε, η βιοπικιλότητα μεταξύ άλλων αυτό είναι το θεματολόγιο που δεν αφορά γενικές αξίες είναι ένα θεματολόγιο που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τα συμφέροντα της Ευρώπης και όπως σας είπα από μια κάποια άποψη του κόσμου. Σε, αυτή, σε αυτό λοιπόν το θεματολόγιο ε, περιμένουμε και την τοποθέτηση των ε, χωρών και γίνεται δουλειά επ' αυτού ε, στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρατε εσείς. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, η Αφρικανική Ένωση ε, συναντιέται στο Κιγκάλι. Ο Ειρηνικός, ε, μεταξύ άλλων, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και είμαι σίγουρος ότι ο παρακατήμενος μου ε, θα εξηγήσει τη θέση των χωρών και αυτή που θα παρουσιαστεί το Μάιο. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τη σημασία της αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς φιλόδοξος, αλλά είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνει υπόψη και κάποια στοιχεία της πραγματικότητας. Αυτό που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία του Κοτονού ήταν ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις τρεις αυτές περιοχές. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το επεξεργαστεί περισσότερο το δεύτερο πάνελ, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι η Αφρικανική Ένωση έχει τη δική της δυναμική και οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αφρική ορίζονται όσον αφορά το στοιχείο της ιδιαιτερότητας ορίζονται διαφορετικά από το θεματολόγιο μας που έχουμε αναπτύξει με την Καραϊβική και με τον Ειρηνικό. Άρα δηλαδή σε αυτό το νέο πλαίσιο είναι απαραίτητο να ενταχθούν ε, τα βασικά συμφέροντα αυτών των τριών περιοχών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βασίζουμε την πρότασή μας ε, στα θεμέλια αλλά και σε πολύ ισχυρούς πυλώνες που κατ' ουσίαν θα συνενώνουν τις ε, διαφορετικές περιοχές, αλλά θα επιτρέπουν και σε εμά ε, και στους εταίρους μας να προβάλλουμε και κοινά και αποκλίνοντα συμφέροντα. Εξάλλου, στο πλαίσιο της πρότασής μας εξετάσαμε και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από την ομάδα των χωρών ΑΚΕ. Αυτό είναι απαραίτητο, κυρίως στην περίπτωση της Αφρικής, όπου η Ευρώπη έχει συμφωνίες σύνδεσης με κάποιες από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπου όμως παράλληλα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συναντηθούμε με την Αφρικανική Πύρο στο σύνολό της, στο Μπιτζάμπ. Είχαμε συνάντηση κορυφής και υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να την παντρέψουμε με δύο διαφορετικές διαφορετικές νομικές καταστάσεις, συμφωνία ε, σύνδεσης με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και την ανάγκη να υπάρξει νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και. Η πρότασή μας λοιπόν εξηγεί ποια ακρίβεια μπορούμε να προχωρήσουμε. Και φτάνω σε ένα θέμα ε, που είναι Αυτό που θέλουμε είναι μια συμφωνία νομικά δεσμευτική. Αυτός είναι ο στόχος των συζητήσεων. Η δική μας η πρόταση είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία έτσι ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε με αυτά που υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου να τα συνδυάσουμε και να τα εντάξουμε στη σχέση μας με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτή τη στιγμή το Κοτονού είναι μια συμφωνία σύνδεσης και αυτό που θέλουμε ως συνέχεια του Κοτονού είναι πάλι μια συμφωνία σύνδεσης ε, που να είναι και νομικά δεσμευτική. Τελευταία παρατήρηση σχετικά με τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κονδύλια αυτό το θέμα δεν καλύπτεται από την σύσταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αυτή τη στιγμή συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Για τον απλούστατο λόγο ότι εξακολουθούμε να εξετάζουμε το επόμενο, ε, την επόμενη πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν όλα πάνε καλά, αυτό θα συζητηθεί στις 2 Μαΐου και εκεί ενδέχεται να προβλέπεται και προβλέπονται κονδύλια για την πολιτική μας. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι σε παράλληλες συζητήσεις που έχουμε θα οργανώσουμε και συζήτηση για το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, άρα δηλαδή και για την επόμενη δέσμη μέτρων οικονομικής ε, βοήθειας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η πρότασή μας συζητιέται στις διαφορετικές ομάδες εργασίας, τα κρατη και όπως σας είπα είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις έχοντας κατά νου ότι θέλουμε εντολή δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου. Αυτό να γίνει ε, το Μάιο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κάτι που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Οι ε, εταίροι μας των χωρών έχουν παρεμφερές ε, χρονοδιάγραμμα και αυτοί μάλλον μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουν πάρει εντολή. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι πραγματεύσει ακριβώς όπως προβλέπεται στη Συμφωνία Κοτώνου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Πράγματι, περίπου τηρήσατε το χρόνο σας. Εντάξει, λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, μια χαρά. Μακάρι να συμβεί και το ίδιο με τον πρέσβη Σιμπουσίβε Μουγκομεζούλου, που είναι πρέσβης της Σουαζιλάνδης και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πρέσβεων των χωρών ΑΚΕ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής ανάπτυξη. είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να σας παρουσιάσω την εισήγησή μου εκ μέρου της Προέδρου της Επιτροπής των Πρέσβειων των χωρών ΑΚΕ. Και θα αρχίσω ευχαριστώντας τους οργανωτές για την ακρόαση αυτή που οργάνωσε η Επιτροπή ε, Ανάπτυξης και κυρίως να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, την ε, κυρία Μακάβαν, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν ε, στην ε, συνεδρίαση αυτή. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της Προέδρους μας, της εξοχώτης της κυρίας Σίλα Σίλι Μοντέιτ από την Τζαμάικα που δεν μπόρεσε να έρθει. Πριν μπω στην ουσία θα ήθελα να συζητήσω λίγο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, νέα συμφωνία και να σας πω ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο, για μια νέα συμφωνία. Κάτι πολύ φιλόδοξο, αλλά και πάντα έτσι ξεκινάμε, με μεγάλη φιλοδοξία. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές ε, εξελίξεις. Οι χώρες μέλη και οι λαοί μας προσβλέπουν ακριβώς αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όλες τους επιθυμίες να ληφθούν υπόψη. Αυτό για μένα αποτελεί σημείο εκκίνησης, να ξέρετε. Και αυτό θα έχω υπόψη μου όσο προχωράμε. Η σημερινή μου παρουσίαση θα αρχίσει με το πλαίσιο των σχέσεων ΑΚΕ Ένωσης και μετά θα ασχοληθώ με τους στόχους μιας νέας συμφωνίας και θα σας μιλήσω για τους πυλώνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως επίσης και για τη δομή των διαπραγματεύσεων. Και στο τέλος θα αναφερθώ στην προπαρασκευαστική διαδικασία ΑΚΕ, όπως ε, και με τους ακρογωνιαίους λίθους που πρέπει να παρουσιαστούν στο τέλος. Λοιπόν, ποιο είναι το πλαίσιο πρώτα απ' όλα. Η αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ των χωρών Αφρικής, Καραβικής και Ειρηνικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ιστορία πολλών δεκαετιών με διάφορα επίπεδα ανάπτυξης, με αλλαγές στις ανάγκες των εταίρων, εξελίχθηκε η σχέση αυτή. Από τότε που υπεγράφει η πρώτη συμφωνία για οντέ 1 μέχρι την πιο πλήρη συμφωνία που είναι αυτή του Κοτονού, η οποία και εκπνέει τον Φεβρουάριο του 2020. Και βάσει του άρθρου 95.4 η ρήτρα αναθεώρησης και επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας αυτής πρέπει να αρχίσει τον Αύγουστο του 2018. Υπό το πνεύμα λοιπόν τη συμφωνία αυτή, που διέπει τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών ε, ΑΚΕ μα φέρνει σε νέε διαπραγματεύσει. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της νέας συμφωνίας. Προβλέπουμε η νέα συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλάβει διάφορες αρχές, στόχους και κατευθυντήριε γραμμές θα πρέπει να ενισχύσει και να βαθύνει περισσότερο την εταιρική σχέση. Θα πρέπει να ενισχύσει την περιφερειακή ολοκλήρωση με την ομάδα ΑΚΕ να λειτουργεί περισσότερο ως ένας αποτελεσματικός παγκόσμιος εταίρος. Τώρα έρχομαι στην δομή. Προετοιμάζοντας τις διαπραγματεύσεις το 104ο Συμβούλιο των χωρών ΑΚΕ που συνεδρίασε πρόσφατα καθόρισε τους εξής στρατηγικούς πυλώνες για μετά το 2020. Πρώτον, εμπόριο, επενδύσεις, βιομηχανοποίηση και υπηρεσίες. Δεύτερον, αναπτυξιακή συνεργασία, τεχνολογία, επιστήμες, καινοτομία και έρευνα. Τρίτον, πολιτικός διάλογος και υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες λοιπόν στους οποίους βασιζόμαστε. Επιπλέον υπάρχουν και κάποιες κατευθυντήριες αρχές πάνω στις οποίες συμφωνήσαμε, που περιλαμβάνουν την διατήρηση και τη ε, συνέχεια που θα δοθεί στο κεκτημένο της ήδη υπάρχουσας εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, να φροντίσουμε ώστε η ομάδα ΑΚΕ να αποτελέσει έναν διακυβερνητικό παράγοντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα, αναγνώριση της επικορικότητας, της πληρωματικότητας και της αναλογικότητας σε σχέση με περιφερειακές και υπηρετικές ομάδες. Έπειτα, να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, οικονομικός για την ανάπτυξη στην ε, συμφωνία. Τώρα προετοιμάζοντας το 105ο Συμβούλιο ΑΚΕ ε, του Μαΐου του 2017, δόθηκε εντολή στην Επιτροπή των Πρέσβεων να δημιουργήσουν μια κεντρική διαπραγματευτική ομάδα και τρεις τεχνικές ομάδες συνολικά που θα στηρίξουν το κεντρικό, την κεντρική ομάδα διαπραγματεύσεων και θα φροντίσει για τη σύνθεση. Η Επιτροπή Πρέσβων λοιπόν τον Οκτώβριο του 2017 ενέκρινε τις κατευθυντήριες αρχές και ε, τα σημεία αναφορά των ε, στοιχείων αυτών. Τη σύνθεση των ε, ομάδων, της κεντρικής διαπραγματευτικής ομάδας και των τριών τεχνικών ομάδων. Η σύνθεση έχει συμπληρωθεί. Λοιπόν, υπάρχει η κεντρική διαπραγματευτική ομάδα η οποία βρίσκεται σε υπουργικό επίπεδο και θα δίνει καθεδρίες γραμμές και υποπτία. Το CNG θα είναι σε επίπεδο πρέσβεων και θα είναι υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις κρίσιμων θεμάτων. Και οι τρεις τεχνικές ομάδες θα είναι υπεύθυνε για διαπραγματεύσεις στους τομείς που η κάθε μία είναι αρμόδια. Προβλέπεται επίσης ότι οι δομές αυτές θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους και αποτελεσματικά να εκπροσωπήσουν τους λαούς των χωρών ΑΚΕ. Όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Τέλος, η προπαρασκευαστική διαδικασία εν ώψη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων πρέπει να ξέρετε ότι συνεχίζονται. Ήδη έχουν αναλυφθεί διάφορες ε, συναντήσεις και πρωτοβουλίες υπάρχει η δήλωση Σαπόπο πρώτα απ' όλα του Δεκεμβρίου του 2012. Υπάρχει επίσης και η δήλωση του Αγκάνη που αποτελεί και τη βάση για την μελλοντική ομάδα. Υπάρχει ομάδα εργασίας σε επίπεδο πρέσβεων για το μέλλον των προοπτικών της ομάδας ΑΚΕ που δίνει παρετέρω κατευθυντήριες γραμμέ. Η ομάδα και επίση έχει αναλάβει διάφορε δραστηριότητε. Έχει κάνει ανάλυση σε βάθο και μελέτε, έχει προετοιμάσει έγγραφα πολιτική που θα δώσουν κατευθύνσει στι διαπραγματεύσει. έχει προχωρήσει αποστολέ σε πρωτεύουσε χωρών και αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υπάρξει και συνομιλίε μη κρατικού φορεί, αλλά και κοινοβουλευτικού. Επιπλέον υπάρχει ειδική επιτροπή πρέσβεων που πρόκειται να ολοκληρώσει τη σύνταξη της διαπραγματευτικής εντολής μέχρι τα τέλη του Απριλίου. Και η έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής της ομάδας ΑΚΕ αναμένεται στο 107ο Συμβούλιο που προβλέπεται για το Μάρτιο του 2018. Η προπαρασκευαστική εργασία χαρακτηρίζεται από πολλές προσπάθειες που είναι όμως συντονισμένες και έτσι το έργο συνεχίζεται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Καρεβικοί και ο Ειρηνικός έχουν ήδη έτοιμες τις τοποθετήσεις τους και το ακούσαμε και πριν. Η Αφρικανική πλευρά έχει επίσης ετοιμάσει τη δικιά της τοποθέτηση, αλλά αναμένεται να εγκριθεί από τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων ε, αφρικανικών χωρών που θα γίνει στο Κιγκάλι, στη Ρουάντα. Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά την αξία της σχέσης των χωρών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο ολοκληρώνεται άλλη μια δεκαετία, εξού και οι χώρες μέλη ΑΚΕ προσβλέπουν σε ανανομένη περίοδο στενών σχέσεων μεταξύ μας και μετά το 2020. Σας ευχαριστώ λοιπόν αυτό το ένδοξο σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευκαιρία που μου δώσατε και σας εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ ε, εξοχότατε. Ακριβή και τηρήσατε και το χρόνο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίε που μας δώσατε. Να περάσουμε τώρα στον τελευταίο μιλητή για αυτό το πρώτο πάνελ, ο Βιβανού Γνασουνού, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ε, των χωρών ε, ΑΚΕ, των σωμάτων χωρών ΑΚΕ, για να κάνει μια ακόμα εισαγωγική παρέμβαση και μετά θα υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, είναι προνόμιο για τη Γραμματεία να σας απευθύνει το λόγο εδώ στην Επιτροπή αλλά μάλιστα να μιλήσει και μετά από την Επιτροπή και τον ε, ε, Αντιπρόεδρο της Ομάδας των Πρέσβεων. Ε, θα μπορούσα να σταθώ σε κάποια πράγματα σε τρία επίπεδα. Καταρχάς να σας πω λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Πώς προσπαθούμε να το κάνουμε και με ποιον προσπαθούμε να το κάνουμε. Και θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω κάποια στοιχεία και ίσως να προσδώσουμε και λίγο σθένος στα όσα προσπαθούμε να κάνουμε από κοινού στα πλαίσια της ανανέωσης της εταιρική σχέσης που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επανέλθω στη βάση τα αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε, διότι και ο πρέσβης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμησαν ότι από το 2011 η ομάδα χωρών ΑΚΕ έχει ξεκινήσει να εξετάζει τις προοπτικές και την προσέγγιση που θα πρέπει να έχει το μέλλον της ε, για μετά το 2020. Αυτό γίνεται σε αρκετά επίπεδα. Ε, ε κορυφώθηκε με τη σύνοδο στην Παπούα ε, το 2016 και ε, εκεί σε πρώτο στάδιο αναγνωρίσαμε ότι πρέπει να αναδιαμορφώσουμε λίγο την προσέγγιση που έχουμε ακολουθήσει και επίσης σε δεύτερο στάδιο ότι θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη αυτή η ομάδα. Είναι μια δήλωση αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων, δεν είναι σε υπουργικό επίπεδο. Να παραμείνει η ομάδα λοιπόν ενωμένη για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε μια νέα δύναμη σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ε, συνεχώς μεταβάλλεται ε, ε, η Επιτροπή αναφέρθηκε στον πολυπολικό κόσμο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απολικός ο κόσμος. Ο καθένας δρά στο επίπεδό του, σε προσωπικό επίπεδο και ε, ενσωματώνει τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζει. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε ε, να προχωρήσουμε. Όταν ε, συστήθηκε η ομάδα το 1975, μόλις είχε γεννηθεί η ομάδα αυτή ε, συστήθηκε το 1975 και το 1975 όταν ε, οι χώρες ΑΚΕ ε, συστήθηκαν σε ομάδα είχαμε μια περιφερειακή ομάδα η οποία ακόμα δεν είχε λάβει συγκεκριμένη μορφή. Ε, συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είχε και μερικές δεκαετίες πίσω της. Οι χώρες ΑΚΕ ήταν ουσιαστικά οι πρώτες χώρες που συνειδητοποίησαν ότι σήμερα ως ομάδα είμαστε, ε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούσαμε. Η σχέση που είχαμε ε, με τις χώρες που μας αποτελούν πρέπει να αλλάξει. Και εκεί ξεκίνησε ο πρώτος προβληματισμό ε, και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερο και να δούμε πώς μπορούμε να ε, συμπληρώσουμε τη σύνθεση της ομάδος. Για μας σήμερα είναι χαρά να γνωρίσουμε ότι σε επίπεδο περιφερειακών ομάδων, για παράδειγμα να πω ότι η CDO e κατάφερε να κάνει αυτά που έκανε στην Κάμπια, κανένα άλλος δεν θα μπορούσε να το καταφέρει ε, από πλευράς Αφρικής και είναι χαρά για μας να λέμε ότι ε, και στην ε, ε, περίοδο μετά την Κοτονού, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε το θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030, αλλά να το κάνουμε βασιζόμενοι, για παράδειγμα, όσον αφορά την Αφρική, στο θεματολόγιο μετά από το 63, γιατί είναι αυτό το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Και τα ερωτήματα που θέτουμε σε επίπεδο ΑΚΕ είναι πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε την όλη διαδικασία. Το πώς θα γίνει περνά καταρχάς από αυτό το διάλογο που επιθυμούμε, που ζητήσαμε και που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε με τις διάφορες ε, ε, χώρες της ομάδος. Ε, και πέρα από τη διαδικασία του προβληματισμού προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να ανανεώσουμε ε, τη λεγόμενη συμφωνία του Georgetown που είναι η δική μας συνθήκη, δεν ξέρω αν είναι η συνθήκη της Λισαβόνα ή του Μάσρι, αλλά είναι η, συνθή... η συνθηκη ιδρυση τη ομάδας Κορονακέ και προσπαθούμε να την αναδιατυπώσουμε για να δώσουμε νέο ρόλο ε, στα μέλη της ομάδος. Γιατί η ομάδα των χωρών ΑΚΕ αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που ε, φαίνονται διάσπαρτοι. Παραδείγματο χάρη, μικρέ χώρες ε, νησιωτικές οι οποίες αναπτύσσονται. Τέτοια μικρά νησιωτικά κράτη έχουμε 37. Τα 36 είναι στην Αφρική. Μήπως τα συμφέροντα αυτών των 37 χρονο, ε, χωρών ή τουλάχιστον αυτών που βρίσκονται στην Αφρική να έχουμε ένα περιβάλλον που έχουμε περισσότερες χώρες που ε, μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα και να μην προσπαθούν να μιμηθούν το θεματολόγιο της Αφρικανικής Ένωσης. Ε, σε επίπεδο Αφρικανικής Ένωσης θα μιλήσουμε, ε, για παράδειγμα, για υποδομές οι οποίες δεν έχουν σχέση με τις υποδομές που χρειάζονται αυτά τα νησιωτικά κράτη. Σε επίπεδο χωρών ΑΚΕ θα μπορούμε να τα δούμε στις δικές μας τις διαστάσεις, διότι η ομάδα των χωρών των νησιωτικών θα μπορέσει να εργαστεί με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο για να δούμε πώς ε, οι χώρες αυτές ε, και θα έχουν τρόπους συνεργασίας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Προηγουμένως αναφερθήκαμε στις υπερπόντιες ε, περιοχές και εδάφη. Αντίστοιχα, ίσως πρόκειται για συλλογική αποτυχία. Δεν καταφέραμε να ε, προχωρήσουμε τη συμμαχία που θα μπορούσαμε να έχουμε με τις υπερπόντες περιοχές και δάφη. Παρ' όλα αυτά έχουμε την ίδια δομή με αυτές τις χώρες, γιατί οι χώρες αυτές έχουν δύο τμήματα, μία πηγαίνουν προς τις χωρές ΑΚΕ και μία προς τις υπερπόντες περιοχές και δάφη τελικά. Ε, και παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε, αποτύχαμε συλλογικά ε, και η γεωγραφική εγκύτητα με αυτές τις περιοχές, με κάποιες από τις χώρες μας, ε, μας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Πέραν του Brexit ή όχι, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας και να μπορέσουμε να βρούμε και μέσα συνεργασία επιπλέον που θα μας βοηθήσουν για τα θέματα αυτά. Το θέμα λοιπόν του ποιος ε, και όχι μόνο με ποιον θα συνεργαστούμε έχει σημασία. Τα κράτη-μέλη των χωρών και συμμετέχουν ε, στα Ηνωμένα Έθνη, οι αφρικανικές χώρες συμμετέχουν και στην Αφρικανική Ένωση και πρέπει να τα δούμε όλα αυτά κάθετα και να μην τα βλέπουμε απλώς ε, συγκυριακά. Ε, η κάθε χώρα θα πρέπει να βλέπει πώς μπορεί να καθορίσει τη στρατηγική της και πώς μπορεί να το γίνει στο κατάλληλο επίπεδο αυτό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα που πρέπει να έχει κάθε χώρα σε κάθε σύνθεση. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα θα ήταν ίσως να πούμε ότι δεν μπορούμε ως περιφερειακές ομάδες να συνεργαστούμε με τις χώρε ΑΚΕ γιατί ε, είναι σαν να μπαίνουμε στα, στη μέση της δουλειά των χωρών ΑΚΕ και θα κάνουμε τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό γιατί δεν έγινε ποτέ και έχουμε για παράδειγμα αυτά που έχουμε στις συμφωνίες ε, Κοτονού, ε, τη διευκόλυνση για την ειρήνη. Εν έχει υλοποιηθεί από την Αφρικανική Ένωση, γιατί η Αφρικανική Ένωση είναι αυτή η οποία έχει τη δυνατότητα και την εντολή να δράσει όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια στι περιοχέ μα. Υπάρχει επίση η δουλειά που γίνεται στον ειρηνικό για κάποια προϊόντα. Έχουμε συνεργασία με τις χώρες αυτές για να τα προχωρήσουν σω λοιπόν αυτή η ποικιλομορφία σε γεωγραφικό επίπεδο θα μπορούσε να ενισχυθεί. Δεν γίνεται αυτό πλήρω σήμερα και να μπορέσουμε ίσως να τα καθορίσουμε αυτά όταν θα καθορίσουμε του στόχου μα και να περιλαμβάνουν όχι μόνο τι χώρε μα, αλλά και χώρε εταίρου, ε, χώρε συνδεδεμένε, ε, Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την ε, Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωση Κορονακέ, αλλά πρέπει να δούμε και πώ θα συνδεθούμε με άλλε χώρε, οι οποίε μαζί μα θα μπορέσουν να προχωρήσουν και κάποιε πολιτικέ και πώς μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη επιρροή και μεγαλύτερο αντίκτυπο με χώρες που, με τις οποίες συνορεύουμε και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μαζί τους περισσότερο. Και αν όντω θέλουμε οι πολιτικές μας να αποκτήσουν κάποια αξία, θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια παρουσίαση η οποία είναι απόλυτα ε, εύστοχη και έχουμε ένα τέταρτο 20 λεπτά για να συζητήσουμε αν παρατείνω κατά 10 λεπτά το πρώτο τμήμα, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στα μέλη, στους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες και που έχουν διάθεση να λάβουν το λόγο φυσικά. Αν μπορέσετε σας παρακαλώ να είστε λίγο συγκεκριμένοι, Σάρλ, ξέρω ότι δεν είναι και το στοιχείο σου, αλλά κάνε μια προσπάθεια ναι, για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους τους αδέλφους που θα θέλεις να πάρουν το λόγο. Ο Σάρλ Γκέρενς, η Σεσίλ Κιέγγε. Άλλος κανείς. Ξεκινάμε λοιπόν. Σάρλ, πόσο χρόνο μου δίνεις. 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό. Τι θα πω σε 1,5 λεπτό. πέντε παρατηρήσεις μετά από την εισαγωγικές ε, αυτές τις παρεμβάσεις που ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχάς, σήμερα έχουμε και άλλους παράγοντες ε, στο τομέα της συνεργασίας μας, παράγοντες οι οποίοι ορισμένες φορές έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, για παράδειγμα την Κίνα. Ε, που έχουμε μεγάλες διαφορές επίσης όσον αφορά την αντίληψή τους για τη διακυβέρνηση, την ε, διεθνή συνεργασία για το εμπόριο, τις διεθνείς σχέσεις ε, και το ρόλο που έχουμε να διαδραματίσουμε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι ο κύριος Κούναρ πολύ σωστά αναφέρθηκε σε μια διεθνή συνεργασία και να υπενθυμίσουμε ότι στα Ηνωμένα Έθνη έχουμε την πλειοψηφία είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουμε και νέο, δύο νέους παράγοντες οι οποίοι ε, είναι εγγεγραμμένοι στη Συμφωνία της Κοτονού. Ε, ο ιδιωτικό τομέα και η κοινωνία των πολιτών. Δεν έχουμε κάνει αρκετή δουλειά από αυτού, πρέπει να τα ενισχύσουμε όλα αυτά. Και τρίτον, όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών αξιών, να πω ότι και εδώ υπάρχει μια πτώση, διότι κάποιες χώρες και κάποια κράτη-μέλη, ΑΚΕ, αντιστάθηκαν ε, την ε, ε, προστασία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται στα μετώπιστεν βεβαίω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο ο οποίο θα λαδώσει τη μηχανή. Αν λάβουμε υπόψη μα ε, τι δεσμεύσει που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε αυτέ, δεν θα πρέπει να αποτελούν πολύ σημαντικό πρόβλημα, διότι συμφωνούν, για παράδειγμα, να ε, διπλασιαστεί η βοήθεια για την ανάπτυξη μέχρι το 2030, λαμβάνοντα υπόψη και τον πληθωρισμό και την παραγωγή και την αύξηση του ΑΕΠ. Ε, δεν θα είναι πρόβλημα λοιπόν αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει μια πτυχή την οποία δεν τονίζουμε αρκετά, η πολιτιστική πτυχή. Έχουμε μια εγκύτητα με τις χώρες ΑΚΕ, ε, που δεν έχει κανένας άλλος ε, μεγάλος παράγον στον κόσμο, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία. Η αγγλική γλώσσα ε, μιλιέται περισσότερο στις χώρες αυτές από ότι στην Αγγλία. Τα γαλλικά, για παράδειγμα στο Κονγκό, έχει περισσότερους γαλλόφωνους από τη Γαλλία. Και όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε αρκετά, δεν γνωρίζουμε τον πολιτισμό των χωρών αυτών. Σε πολιτιστικό επίπεδο λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχω πολλά ακόμα να πω, αλλά επειδή ο κύριος Έγγελ ε, ε ασκεί πολιτική λιπτότητα, ε, θα σταματήσω εδώ. Έτσι κι ήμουν και ως το Λουξεμβούργο όταν ψηφίστηκε ο νόμος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω τελικά όπως σας είπα. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συζητητές ε, για το πλαίσιο που σκιαγράφησαν όσον αφορά την περίοδο μετά το Κοτονού. Τους ευχαριστώ και για τις προτάσεις που κατέθεσαν. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν άκουσα να λέγονται πολλά για το μέλλον της ισομερούς κοινοβουλευτικής συνέλευσης και από τις δύο πλευρές. Ε, θα ήθελα να ξέρω τι θα γίνει ποιο είναι το σχέδιο αυτής της ισομερούς κοινοβουλευτικής συνέλευσης, δηλαδή πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση και ε, πώς ακριβώς εσείς μπορέσατε να φτάσετε στο να σχεδιάζετε την επόμενη στρατηγική για αυτή τη συνέλευση που είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αν σήμερα μιλάμε για τον πολιτικό διάλογο πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι ο πολιτικός διάλογος ξεκινάει ακριβώς μέσα σε αυτή τη συνέλευση. Ως εκ τούτου η δυνατότητα να ενισχυθεί η συνέλευση αυτή η δυνατότητα είναι κάτι που πρέπει να υπόψη. Ε, το δεύτερο θέμα που το έθιξε και ο συνάδελφος Γκέρενς είναι η κοινωνία των πολιτών. Ε, μετά το Κοτονού είναι η κοινωνία των πολιτών τώρα σε αυτή τη διαδρομή πώς ακριβώς εμπλέκεται η κοινωνία των πολιτών ε, από τώρα μέχρι και την περίοδο μετά το Κοτονού. Και εμείς ευχαριστούμε. Αν δεν... Α, η Λίντα. Εγώ τα ήθελα απλά να ερωτήσω τους ομιλητές, κυρίως τον Κούν, να τον ρωτήσω, τον κύριο Κούνχαρτ μάλλον, όχι τον Κούν, τον Ντονς, το θέμα της Βόρειας Αφρικής. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά στην πράξη ίσως ε, να πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί πιστεύαμε ότι χώρισα και αυτό συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση και να μας πούνε και οι φίλοι μας από τις χώρες και τι πιστεύουν εκείνοι. Το να ανοίξουν, να ανοίξει η συνεργασία, πώς θα λειτουργήσει αυτό πρακτικά ε, κάτω από το δικό σας πρίσμα. Στο δεύτερο τμήμα θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο ε, γιατί έχει ε, οριστεί ως καθοριστικό στοιχείο για τη συνεργασία. Η πιθανή πρόταση της Κομισιόν για το Μάιο είναι αυτό το Ταμείο να ενταχθεί στον προεπλογισμό, να υπάρχει δηλαδή ένα και μόνο Ταμείο για όλες τις εξωτερικές δράσεις. Αυτό μάλλον θα είναι το αποτέλεσμα δεν ξέρω εσείς ε, πώς το φαντάζεστε αυτό, πώς θα λειτουργεί αυτό πρακτικά, διότι οι εταίροι μας ε, από τις χώρες ΑΚΕ έχουν συνηθίσει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για κάθε χώρα, μία μακροχρόνια χρηματοδότηση. Η Κομισιόν το έχει σκεφτεί αυτό και να μας πούνε και οι εταίροι μας από τις χώρες ΑΚΕ ε, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Ε, μας λένε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ε, για να προχωρήσουμε, ε, κυρίως όσο προχωράνε και οι διαπραγματεύσεις. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Πριν λοιπόν επανέλθω στους ομιλητές, θα ήθελα να καλέσω την Κριστίν Ντεπερόν από την, Ευρωπαϊκή, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μιλήσει και εκείνη να μας ε, ενημερώσει και μετά θα επανέλθουμε στους ομιλητές του πάνελ για να ολοκληρωθεί ο γύρος ε, και θα μείνει και χρόνος για μένα για να παραδώσω στον Νόρμπερτ ε, για το δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη γιατί συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά για τα μετά του Κοτονού. Οπότε δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Κούν Ντούνς. Κάποια σημεία όμως θα ήθελα να θίξω και ένα από αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ότι έχουμε κληρονομήσει από τη Συμφωνία Κότων, που είναι ο πολιτικός διάλογος. Έχουμε σε επίπεδο ΑΚΕ, αναφέρθηκε, αλλά έχουμε και έναν καθημερινό και πιο συχνά είναι σε επίπεδο χωρών, με κάθε χώρα δηλαδή χωριστά. Έχει χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα αυτή όσο μπορούμε και πιστεύουμε ότι σε μια σύγχρονη εταιρική σχέση, μια που μιλάμε για το 2030, για τους στόχους του 2030, νομίζω ότι μπορούμε σε αυτή τη νέα ε, σχέση να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και σε επίπεδο ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο περιφοριακό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο μεταξύ μας και να συζητήσουμε θέματα που έχουν ε, να κάνουν με τις ανησυχίες της κάθε χώρας. Έχουμε συνεργαστεί έτσι για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και καταλήξαμε σε σημαντικές τοποθετήσεις που έχουν αλλάξει πράγματα, αλλά Υπάρχουν και άλλοι τομείς, η μετανάστευση, και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα μαζί, αλλά σίγουρα και άλλα περιβάλλον, χρηματοδότηση της ανάπτυξης κλπ. κλπ. Συνεπώς, ο στόχος να υπάρξουν πολυεπίπεδες σχέσεις θα ενισχύσει την εταιρική μας σχέση. Και μια που πρόκειται για μια εταιρική σχέση σύγχρονη, που βασίζεται στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει εκατέρωθεν, όταν έχουμε πολιτικό διάλογο, δεν θα πρέπει να συζητάμε μόνο την εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες, αλλά να συζητάμε θέματα που μας απασχολούν αμοιβαία και έχουν να κάνουν με τη διεθνή σκηνή. Να συζητήσουμε και πράγματα που ανησυχούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα που ανησυχούν τους εταίρους των χωρών και και έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την εταιρική σχέση και πώς εμείς την αντιλαμβανόμαστε, ο Κουν περιέγραψε πώς βλέπουμε εμείς τις νέες βάσεις για αυτήν την σύγχρονη συμφωνία. Οι προτάσεις που έχουν γίνει για τους περιφερειακούς πυλώνες έχουν σαν στόχο να δούμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά στο κατάλληλο επίπεδο. Όσον αφορά την εταιρική σχέση με την Αφρική, εκεί έχουμε μια εταιρική σχέση για το περιβάλλον συνολικά με την Αφρικανική Ήπειρο. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η εταιρική σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο, με την Βόρεια Αφρική να παραμείνει, να παραμείνει δηλαδή αυτή η ιδέα της κοινή απόφασης όπω συμμετέχουν όλοι για θέματα τα οποία αφορούν όλους τους Αφρικανούς εταίρους μας. Όταν πρόκειται βέβαια για την υλοποίηση υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν ε, δομές, υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης κλπ. Αλλά θέλουμε πολιτικά τη συμμετοχή όλων των Αφρικανών εταίρων. Θα σταματήσω όμως εδώ γιατί θα είμαι σύντομη. Ο κύριος Έγκελ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, οπότε μπορώ τώρα να δώσω το λόγο στου, στα μέλη του πάνελ εδώ. Τρία λεπτό καθένας για να απαντήσει στα σχόλια. Και ο καθηγητής Κιούνερτ από ό,τι κατάλαβα θα πάρει το λόγο στο τέλος. Οπότε, να αρχίσω με τον Κουν ή ανάποδα. Ανάποδα. Εντάξει, τότε θα αρχίσουμε από τον Γενικό Γραμματέα ΑΚΕ. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω σε δύο δικές ερωτήσεις και μετά θα βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα. Πώς βλέπουμε εμείς την Νέα Σύμφωνη. Πώς βλέπουμε εμείς τους εκτελεστικούς εταίρους. Εμείς θέλουμε μια εταιρική σχέση που να είναι γεμάτη δυναμισμό. Και ο δυναμισμός αυτός πρέπει να είναι εκτός εκτελεστικών θεσμών επίσης. Γι' αυτό και συζητάμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν χρησιμοποιεί από κοινού θεσμούς, πάντα ad hoc όταν πρόκειται για κοινοβουλευτικέ συναντήσει σε περιφερειακό επίπεδο, λέει ότι πρόκειται για σχέση ad hoc. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η θεσμική σχέση που προτείνεται. Στην πρόταση ΑΚΕ, βέβαια δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε, πρώτα πρέπει να αποφασίσουν οι χώρε. Εμεί ζητήσαμε μελέτε σε διάφορα επίπεδα ακριβώ για την εταιρική σχέση, για την ενίσχυση τη εταιρική σχέση, για να υπάρξουν συστάσει πώ η κοινή μα φιλοδοξία μπορεί να προχωρήσει και τελική αυτή η σχέση να γίνει ακόμα πιο χρήσιμη. Συνεπώς εμπνεόμαστε από αυτήν την ε, μελέτη που ξεκίνησε και στην εντολή θέλουμε να προβλέψουμε ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των μελετών που ζητήσαμε θα αποφανθούμε κιόλα. Το ίδιο και για τη χρηματοδότηση. Ο πρέσβης του Σουαζιλάνδης είπε ποια είναι η διαπραγματευτική εντολή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ένα εργαλείο συνεργασίας. Η τάση είναι συχνά τα μέσα συνεργασίας να τα βάζουμε όλα μαζί σε μία οντότητα. Ακόμα και με θεματικές διαφορές ή περιφερειακή διάσταση. Χρειάζεται όμως προβλεψιμότητα χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και ιδιαιτερότητες. Αυτό πρέπει να παραμείνει, όποια μορφή και αν πάρει τελικά η εντολή αυτή. Οι αρχές πρέπει να διέπουν το όποιο αυτό νέο όργανο, νέα δομή. Τώρα, η επόμενη περίοδος θα είναι μια περίοδος πολύ σημαντική για μας, όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις, αλλά για να τοποθετηθούν και οι χώρες μας στη διεθνή σκηνή. Το θέμα τίθεται. Ακόμα και αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε. Όμως, ό,τι υπάρχει ήδη σήμερα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε σήμερα αν δεν υπήρχε, γιατί η σημερινή δυναμική δεν θα οδηγούσε σε μια τέτοια ομάδα, παρόλο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ύπαρξη της ομάδας τώρα. Και εγώ δεν μιλάω μόνο για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι χώρες του Νότου, σε συνεργασία βέβαια με τον Ειρηνικό και την Καραϊβική που μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ανησυχίες ή τέτοια συμφέροντα με την Αφρική αλλά θέλουν να μας στηρίξουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο ισχύει για το κλίμα που είναι βέβαια μια ανησυχία πολύ πιο έντονη στον Ειρηνικό αλλά η Αφρικανική ομάδα τι λέει. Λέει όχι θέλουμε να σας στηρίξουμε, θέλουμε μαζί να καθορίσουμε το τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον μας και τι θα κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές. Είναι δηλαδή ένας δυναμισμός αυτός που υπάρχει και πάνω στον οποίο πρέπει να βασιστούμε. Μην κάνουμε λάθος. Δεν μπορεί να είμαστε κοντόφθαλμοι. Ό,τι διακυδεύεται τώρα δεν είναι μόνο η εταιρική σχέση, είναι και η ίδια η διατήρηση και η ύπαρξη των λόγων του Νότου που διακυδεύεται εδώ. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε και να προχωρήσουμε έτσι. είναι πάρα πολύ ελκυστικά αυτά που λέτε, γιατί πράγματι αν σήμερα έπρεπε να φτιάξουμε την εταιρική σχέση που υπάρχει ήδη εδώ και δεκαετίε και είναι πολύ καλά δομημένη, θα δυσκολευόμασταν για πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Καλό είναι σήμερα ό,τι προβληματισμό και αν έχουμε, τη δομή αυτή να τη διατηρήσουμε. Παρακαλώ, εσείς τώρα κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουν τεθεί μία σειρά ερωτημάτων και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα όπως τα θυμάμαι. Όσον αφορά το μέλλον ε, της ε, αναπτυξιακής πολιτικής, χτες είχαμε μία συνάντηση των βουλευτών των χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας και σε αυτή την ομάδα εργασίας ε, ε, ορίστηκαν οι αρμοδιότητες. Άρα δηλαδή η όλη ιδέα είναι να υπάρξει ε, ένα πλαίσιο για την κοινοβουλευτική συνέλευση. Και Παράλληλα με αυτό υπάρχει και η δυνατότητα να επαναληφθεί η συμφωνία του Georgetown. Ε, κάποιες ε, περιοχές της Νότιας Αφρικής, ε, ε, εμείς οι συντονιστές από την Σουαζιλάνδη ε, προτείναμε να ενισχυθεί η διάσταση, η κοινοβουλευτική διάσταση. Έτσι λοιπόν αυτό αφορά την περίοδο μετά το 2020. ίσως ε, το επίπεδο της ε, συμμετοχής ε, να είναι περιφερειακό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι σκέψεις που επικρατούν. Όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και πώς μπορεί να προκύψει μια νέα συνεργασία, θέλω να πω ότι υπάρχει ανάγκη για τον πολιτικό διάλογο. Αυτό το χρησιμοποίησαμε, χρησιμοποίησαμε ε, την συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών. Γνωρίζουμε ότι στη δική μας την περιοχή υπήρξε μια συνάντηση τον Νοέμβρη όπου συναντήθηκαν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με εθνικούς ε, παίκτες και εμπλεκόμενους. Το Κοτονού στηρίζει αυτό το ρόλο και πιστεύουμε ότι μετά το 2020 θα πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος. Όσον αφορά το να ανοίξουν τα μία ε, στις χώρες ΑΚΕ, έχει τοποθετηθεί από αυτού η κοινοβουλευτική συνέλευση, αλλά βεβαίως ε, απευθυνόμεθα στους εταίρους μας ε, να εξεργαστούν περιττέρω τον μηχανισμό και το πώς ενδεχομένως θα μπορέσουμε να ενημερωθούμε, να επωφεληθούμε καλύτερα. Και επειδή μιλάμε για αυτά τα θέματα, ε, πρέπει να σας πω, στην ομιλία μου προηγουμένως δεν ανέφερα ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες και από με αυτούς τους τρεις πυλώνες θα ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις ε, όπως ε, ορίστηκαν αυτοί από ε, το Συμβούλιο. Ο πρώτος πυλώνας, οι επενδύσεις και η βιομηχανοποίηση, αφορά στην συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει ότι ο ιδιωτικό τομέας, τα ΣΔΙΤ, ε, είναι μεγάλη σημασία και θεωρούμε ότι χαράσσονται πολιτικές στις χώρες ΑΚΕ για να διασφαλίσουμε την ελκυστικότητα για να μπορέσουμε τις ε, ε, ξένες δημόσιες επενδύσεις να τις κατευθύνουμε στα δικά μας τα κράτη-μέλη. Ε, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα συνεχιστεί. Και όταν μιλήσατε για τον πολιτικό διάλογο, προφανώς εμείς ως κράτη-μέλη συμφωνούμε, θέλουμε να ξεφύγουμε από το να λαμβάνει ένα ακόμα μία μονομερή προσέγγιση σε τέτοιου είδους θέματα. Θέλουμε ε, η όλη η εικόνα του Κοτονού να παραμείνει ζωντανή. Αναφέρθηκα σε θέματα τα οποία αφορούν πολλές χώρες ε, και όπως παραδείγματο χάρη ε, νομοθετική φορολογία που δεν έχει σχέση με τις εταιρείε, μη εταιρική δηλαδή φορολογία. Ε, οι εταίροι μπορούν να συζητήσουν από αυτού του θέματος. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος για να αξιολογήσουμε την πρόοδο αυτών των συζητήσεων πριν όλα αυτά δρομολογηθούν και ενταχθούν μάλλον καλυφθούν από το άρθρο 96, συσχετιστούν με το άρθρο 96. Πράγματι τον χρειαζόμαστε τον πολιτικό διάλογο και ε, πρέπει να ενισχυθεί αυτός για να μην υπάρχουν ε, μαύρες λίστες, λίστες ε, ανεπιθύμητων. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί να αμφισβήτηση. Um, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κούνς, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, κοινή με κοινοβουλευτική συνέλευση και την κοινωνία των πολιτών. Η προσέγγιση που έχουμε είναι η εξής. Ε, να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε ως κινητήρια δύναμη το πολιτικό στοιχείο. Αυτό λοιπόν σημαίνει όχι μόνο όταν συναντιούνται οι υπουργοί, αλλά επίσης όλα αυτά σημαίνουν και όταν συναντούνται οι βουλευτές και όταν συναντιόνται οι κοινωνίες των πολιτών. Σε αυτή τη νέα προσέγγιση θα γίνουν πολλά περισσότερα, δηλαδή θα μετακινηθεί λιγάκι το κέντρο βάρους ε, στους περιφερειακούς πυλώνες. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η κοινοβουλευτική διάσταση, η διάσταση της κοινωνίας των πολιτών να ακολουθήσουν και έτσι να μπορεί κανείς ε, και να συνεισφέρει και να ελέγχει. Όταν θα υπάρχουν ε, ε, υπουργικέ συναντήσεις σε επίπεδο περιφέρειας Καραβικής, Ειρηνικού, ε, Αφρικής, αυτά να ακολουθούνται και με παρεμφερή δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά την, τις χώρες ΑΚΕ Εκεί ε, εντάσσονται οι βασικές μας δεσμεύσεις και όπως πολλοί από εσά είπατε το βασικό θέμα είναι το διεθνές θεματολόγιο. Δηλαδή ποια είναι τα θέματα εκείνα όπου 28, σύντομα 27, συν οι χώρες ΑΚΕ που ακριβώς ε, συμπίπτουν οι απόψεις μας, συγκλίνουν και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το διεθνές ε, θεματολόγιο. Εκεί πρέπει να συναντηθούμε για να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το θεματολόγιο. Παράδειγμα, COP21, αλλά υπάρχουν ε, και πάρα πολλά άλλα θέματα. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο ε, συναντήσεις επίπεδο όπως η COP21, να είναι και άλλου είδους συναντήσεις ε, όπου οι αριθμοί μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Για μας λοιπόν είναι σημαντικό το ότι συγκλίνουν οι απόψεις των θεσμών όσον αφορά την ουσία της συζήτησης. Για τη Βόρεια Αφρική, ερώτηση της Λίντα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα είναι αρκετά ευθύς. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνίες σύνδεσης με χώρες Βόρειας Αφρικής το νέο πλαίσιο, η νέα συμφωνία Κοτονού, θα, αν πάνε όλα καλά, θα δημιουργήσει μια συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ΑΚΕ από την προοπτική της ε, Αφρική σημαίνει ότι και οι υποσαχάρες χώρες και αυτές μπαίνουν σε νομικά δεσμευτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι δύο πλευρές ε, πρέπει να συγκλίνουν, να συναντηθούν κάπου, δηλαδή να υπάρχουν συναντήσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση, το σύνολο των χωρών της Αφρικής. Πώς θα γίνει, όπως γίνεται και τώρα. Δηλαδή πολιτικά θα ε, οργανώνουμε συναντήσεις κορυφής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση και οι ποσαχάρες χώρες και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής αλλά και η Ευρωπαϊκή όλοι συμμετέχουν στη συζήτηση. Το ίδιο θα κάνουμε και σε υπουργικό επίπεδο. Εκεί θα λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις με όλα τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης. Και αν χρειαστεί κάποιες από αυτές τις συμφωνίες να στηριχτούν με νομικά πλαίσια, αυτό θα γίνεται μέσα από τα συμβούλια σύνδεσης. Στην περίπτωση των χωρών της Βόρειας Αφρικής έχουμε ε, δημιουργήσει τις ε, συμφωνίες σύνδεσης και για τις υποσαχάρες χώρες ε, Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποσαχάριων χωρών. Θα μπορούν κατ' ουσίαν όλοι να συναντιόνται την ίδια μέρα, άρα δηλαδή έχουμε ένα μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα έχετε δει το House of Cards και θέλω όμως να σας πω ότι οι συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο συνεχίζονται. Τώρα κατά πόσον θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό το αναπτυξιακό ταμείο ή όχι, δεν έχει σημασία. Θα υπάρχουν τα κονδύλια και ακόμα και αν υπάρχει ένα νέο γεωγραφικό εργαλείο, ένας τέτοιος μηχανισμός, σημασία θα έχει να εντοπιστούν κάποια κονδύλια για μια συγκεκριμένη ομάδα κρατών. Δεν είναι δηλαδή ε, πολλά κονδύλια που απλά θα περιμένουν. Το θέμα είναι να γίνουν αυτές οι προσημειώσεις ακριβώς για να προβλέπονται κονδύλια για συγκεκριμένες ομάδες χωρών που είναι ε, πολύ σημαντικές ε, για, τις, ε, γιατί είναι χώρες λιγότερο αναπτυγμένες ή γιατί είναι εταίροι μας σε χώρες ΑΚΕ. Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Και για να ολοκληρώσουμε το όλο θέμα, πάμε στον καθηγητή κύριο Κιούνχατ, ο οποίος με έχει διαβεβαιώσει ότι προτίθεται να μας κάνει μία μικρή ανακεφαλαίωση και, και περίληψη των όσων ελέγχθησαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πράγματι τονίσατε κάποια από τα θέματα που ανέφερα ε, γι' αυτό και εγώ ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος θα κάνω έτσι μια ανακεφαλαίωση ε, θέλω να πω όλα αυτά αντικατοπτρίζονται με το ρητό που λέει η επιτυχία του μάγειρα φαίνεται από τον τρόπο ή από το φαγητό, από το πώς καταναλώνεται το φαγητό. Θέλω να πω ότι Όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική, είμαι λιγάκι επιφυλακτικός. Βόρεια δεν είναι μόνο γεωγραφικό το θέμα. Ε, το θέμα είναι και ότι δεν υπάρχει εκεί περιφερειακή ολοκλήρωση συνεχίζονται πάρα πολλές εντάσεις σε πολλές από αυτές τις χώρες. Υπάρχει για τη Συρία έλλειψη προοπτικής, ειρήνευσης στην περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι αυτό που είπε ο κύριος ε, Ντόνς. Ε, δεν ξέρω αν αυτό βέβαια είναι και το πιο δημοφιλές. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, επιτέψτε μου να τονίσω αυτά που μόλις ελέγχθησαν, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων. Νομίζω ότι το βασικότερο για την επιτυχία, αλλά και για το πώς το, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται μία μελλοντική συμφωνία, ε, το βασικότερο απ' όλα είναι να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής μέσα από την πρόοδο και αυτό επίσης να το πιστεύουν και οι Ευρωπαίοι. Να υπάρξουν επίσης θέσεις απασχόλησης, επενδύσεις, ε, να έχει κανείς περισσότερες ευκαιρίες ε, στη ζωή του. Στο μέλλον με μη διπλωματικό τρόπο είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι αντιφάσεις της ατελούς παγκοσμιοποίησης. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όσο βλέπουμε περισσότερη μετανάστευση, τόσο περισσότερο ε, θα βλέπουμε πρόοδο στον Νότο. Και φτάνω στο δεύτερο θέμα, στην κοινωνία των πολιτών. Δεν πρόκειται μόνο για τον πολιτισμό γενικά, πρόκειται για τον πολιτικό πολιτισμό, ένας νέος τρόπος ε, να συνενωθούν οι κοινωνίες όπου ε, βιώνουμε την αποαπικιοκρατικοποίηση του νεοκολονιαλισμού, της νεοαπικιοκρατίας. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο όχι μόνο για την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο για τους ε, παραδοσιακούς ε, παίκτες. Έχουμε μια νέα κατάσταση και για πάρα πολλούς άλλους ε, για πολλές επαγγελματικές ομάδες που κατά κανόνα δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσα από το θεματολόγιο βορρά-νότου. Όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο που θα χαράξει νέα συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ. Και αυτά θα προσθέσουν αξία και στις δύο πλευρές και φτάνω τώρα στην τρίτη μου παρατήρηση και μετά από αυτά που ακούσαμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αυτά ε, θα δώσουν σημασία στη μελλοντική συμφωνία, η οποία μπορεί να είναι ένα εργαλείο ε, για πρόοδο ε, και για να προχωρήσει η πολυμέρεια σε μια εποχή ε, όπου η ε, πολυμέρεια αυτή την εποχή σε ολόκληρο τον κόσμο δέχεται πιέσεις. Νομίζω ότι είναι ένας μηχανισμός για να προχωρήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι με την ατελή παγκοσμιοποίηση, όπως την αποκαλώ. Βρίσκεται μπροστά μας ε, και η λειτουργία αυτής της νέας συμφωνίας πρέπει να είναι αποτελεσματική γιατί έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσουμε αυτά τα οποία επεξεργάζεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Ε, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νόμπετ Νόιζα για να ακολουθήσει το δεύτερο πάνελ. Έχουμε λιγάκι καθυστερήσει αλλά θα καλύψουμε το χρόνο που χάσαμε. Ε, Καλησπέρα σας. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Ξέρετε πρέπει να τελειώσουμε στις 5. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους σε αυτό το δεύτερο πάνελ. θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την διαδικασία της περιφερειοποίησης των εταιρικών σχέσεων και πώς μπορούμε μια εταιρική σχέση να την μετατρέψουμε σε μια πραγματική εταιρική σχέση πολλών εταίρων, πώς όλα αυτά μπορούν να γίνουν συμπεριλαμβάνοντας ε, τις ε, τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών. Ξεκινάμε με μια ακαδημαϊκή παρουσίαση του κυρίου Μαουρίτσιο Καρμπόνε, καθηγητή διεθνών σχέσεων και ανάπτυξης ε, στο Πανεπιστήμιο της γλασκόπης. Θα ακολουθήσει ο κύριος Μοχάμπετ Ιγκουα Όφλε, στέλεχος ε, της Αφρικανικής Ένωσης, ε, της μόνιμης αντιπροσωπείας Αφρικανικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσει μετά ο κύριος Jean-Pierre Μπάση, Γενικός ε, Γραμματέας των Ενωμένων Πόλεων και των τοπικών κυβερνήσεων της Αφρικής. Και στο τέλος Καρίν Σοχέ, Πρόεδρος της Concord, Ομάδας Εργασίας των Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ. Επτά λεπτά έχει ο κάθε ομιλητής. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε να ε, κρατηθείτε σε αυτό το χρόνο για να μπορούν και οι συνάδελφοι να σας κάνουν ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Okay, so... Λοιπόν, For an academic it's not easy to talk in... Για έναν πανεπιστημιακό δεν είναι εύκολο να μιλήσει σε 7 λεπτά, αλλά να σας κάνω μια αποκάλυψη καταρχάς. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης με ένα project το οποίο έχει τίτλο «Αναδιαμορφώνοντας τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕΝ», αλλά σαν καλός Ιταλός δεν μπορεί μόνο η κυρία Μογκερίνη να έχει δύο ιδιότητε, Έχω κι εγώ δύο ιδιότητε. Είμαι σύμβουλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τα τελευταία δύο χρόνια και ε, το λέω αυτό για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Σήμερα θα μιλήσω όμως ε, σε προσωπική βάση τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπής. Μόνο ε, ω πανεπιστημιακό στο Πανεπιστήμιο τη Γλασκόβη ομιλώ. Δύο πράγματα έχω να πω. Είναι πολύ δύσκολο να πω τα πάντα σε 7 λεπτά. Μου ζητήθηκε να κάνω μία σύντομη εισαγωγή για τη η περιφερειακή διάσταση, την περιφερειοποίηση. Ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των δύο συστατικών στοιχείων της ε, νέας συμφωνίας. Αφενός υπάρχει μια απόπειρα να παραμείνει το τμήμα του κεκτημένου υπό τη σκέπη μια σειράς από βασικούς στόχους και ε, ένα τμήμα διεθνούς συνεργασίας ε, που είναι πολύ σημαντικό και δεν υπήρχε προηγουμένω, διότι όπως γνωρίζετε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών ΑΚΕ δεν ε, φτιάχτηκε για τη διεθνή συνεργασία πέραν της συνεργασίας μεταξύ των δύο. Και το δεύτερο σκέλος είναι αυτοί οι τρεις πυλώνες. Υπάρχει ένα όριο συνήθως όταν μιλάει ο κόσμος. Υπάρχει μια παρανόηση για την έννοια της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της περιφερειοποίησης. Ε, ήθελα να σας κάνω μια μακρά παρέμβαση για το τι σημαίνει αυτός ο όρος και πιο συγκεκριμένα αυτή η ιδέα της περιφερειοποίησης που είναι μια μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας σε ε, γεωγραφικά περιορισμένη κλίμακα και υπό μία έννοια ε, η περιφερειοποίηση είναι ένα υποσύνολο ε, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ε, η περιφερειοποίηση, να μην συγχαίουμε τους δύο όρους regionalism και regionalization, είναι μια διαδικασία εντός μιας γεωγραφικής περιοχής. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ο ένας όρος στη θέση του άλλου, αλλά δεν είναι το ένα και το αυτό. Και υπάρχει και ένας τρίτος όρος που αναφέρεται στις συζητήσεις που είναι η περιφερειακή τάξη. Η περιφερειακή τάξη, regional order, είναι ένα επίπεδο για διακυβερνητέ, διακρατικές σχέσεις σε μια περιοχή που μπορεί να περιλαμβάνουν ή να μην περιλαμβάνουν ε, θεσμική ε, διακυβερνητική συνεργασία. Και ε, κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι οι διάφορες μορφές ε, περιφερειακού στοιχείου. Ε, μία μορφή είναι ο πολιτικός, το πολιτικό περιφερειακό στοιχείο που αναφέρεται σε θεσμούς των οποίων ο πρωταρχικός ρόλος είναι να προωθήσουν μια αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και να ενισχύσουν τη φωνή μιας ομάδας χωρών σε πολυμερείς οργανισμούς ή ε, πιο γενικά στις ε, παγκόσμιες υποθέσεις. Ο, η πολιτική περιφερειακή διάσταση, αντί να επιβάλλει ε, περιορισμού στην εθνική αυτονομία, μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μπορεί να ενισχύσει το ρόλο και να μεγενθύνει τη φωνή χωρών στις διεθνείς σχέσεις. Ε, υπ' αυτή την έννοια, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Αφρικανική Ένωση είναι μια απόπειρα προς αυτή την κατάσταση. Η δεύτερη μορφή περιφερειακής διάστασης είναι η λειτουργική περιφερειακή διάσταση. Και η λειτουργική περιφερειακή διάσταση περιλαμβάνει μια κάποια διακρατική συνεργασία ε, σε συγκεκριμένα θέματα. Και αυτό ε, μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι μεταφορές οι οποίες ε, θεωρούνται ότι είναι ουσιαστικό πρόβλημα, για παράδειγμα, για την υποσαχάρη Αφρική. Υπ' αυτή την έννοια, η λειτουργική ολοκλήρωση δεν περιορίζει τα κράτη-μέλη στην αυτονομία τους και στην πραγματικότητα παρέχει μία σειρά από ωφέλη στα κράτη-μέλη. Γιατί δημιουργούνται συγκεκριμένα έργα υποδομών και προσελκύονται κονδύλια από εξωτερικούς δωρητές. Υπάρχει και μια τρίτη μορφή περιφερειακής διάστασης, είναι η οικονομική περιφερειακή διάσταση. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο επιβάλλει μια σειρά από περιορισμού στα κράτη-μέλη και αυτές είναι οι μορφές ε, οικονομικής περιφερειακής διάσταση μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές. Άρση φραγμών, ροή αγαθών και υπηρεσιών, μετανάστευση, ροή κεφαλαίων. Ε, πρόκειτο να σας πω μια ιστορία για την εξέλιξη της περιφερειακής διάστασης στην Αφρική, αλλά δεν έχουμε αρκετό χρόνο και έχουμε δει διάφορα κύματα περιφερειακής διάστασης τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα πρώτο κύμα το οποίο ήταν περισσότερο διακυβερνητικό και στο οποίο η οργάνωση της Αφρικανικής Ένωσης ανέλαβε τα ενία στις σχέσεις μεταξύ τμήματων της Αφρικανικής Ένωσης που βασίζονταν κυρίως σε σχέσεις μεταξύ κυβερνήσεων. Και αυτή είναι η συζήτηση που βλέπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια συζήτηση. Η δεύτερη κατηγορία, το δεύτερο κύμα μάλλον περιφερειακής διάστασης που προέκυψε όταν ε, το 2002 συστήθηκε η Αφρικανική Ένωση, είναι πιο πολύ ένας υπερεθνικός θεσμός. Δηλαδή υπάρχει μια απόπειρα να εχωρίσουμε εξουσίες σε κάποια θεσμικά όργανα, υπερεθνικά θεσμικά όργανα, τα οποία συστήθηκαν και υπάρχει και μία απόπειρα να καθορίσουμε πρότυπα για ανθρώπινα δικαιώματα, να καθορίσουμε μία σειρά από κανόνες. Και Το πρόβλημα με την ε, εξέλιξη του, ε, της περιφερειακής διάστασης στην ε, Αφρική είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να λύσει τις σχέσεις μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης Αφενών και ε, του ΡΕΚΣ αφετέρου. Δηλαδή, ε, πολλοί θεωρούν ότι τα ΡΕΚΣ είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο, αλλά πάντα μπορεί να γίνει μια σαφής διάκριση, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ε, της απόδοσης των διαφόρων περιφερειακών οργανώσεων στην Υποσαχάρη Αφρική. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπει σε αυτές τις περιφερειακές οργανώσεις να λειτουργήσουν όπως θέλαμε να λειτουργήσουν είναι ότι δεν υπάρχει σύγκληση μεταξύ των περιφερειακών συμβουλίων. Κάποια φαίνεται να έχουν εγκρίνει μια προσέγγιση προς την ολοκλήρωση που βασίζεται και εδώ σας παραθέτω σε προθεσμίες και μετά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ε, κάποιοι έχουν προχωρήσει σε διάφορα συστατικά στοιχεία, για παράδειγμα ελευθερία κεφαλαίων, αγαθών, ε, κινητικότητα κλπ. Κάτι ακόμα και σε ένα λεπτό τελειώνω είναι ότι η σύσταση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου υποτίθεται ότι θα δημιουργούσε ενδοπεριφερειακό εμπόριο. Και αυτό δεν έχει συμβεί. Ε, μάλιστα τα περιφερειακά συμβούλια δεν έχουν αυξήσει καθόλου το ενδοπεριφερειακό εμπόριο. Το ενδοπεριφερειακό εμπόριο στην Αφρική είναι το μικρότερο στον κόσμο, είναι το 12% του συνολικού εμπαρίου σε σχέση με 20% στην Ασία και 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος υπάρχει και η έλλειψη εναρμόνισης και συντονισμού μεταξύ των περιφερειακών συμβουλίων ε, μεταξύ τους και ε, στις σχέσεις με την Αφρικανική Ένωση. Για την Αφρικανική Ένωση, με άλλα λόγια, τι είναι αυτά τα περιφερειακά συμβούλια. Είναι πυλώνες της Αφρικανικής Ένωσης ή είναι πιο αυτόνομες δομές. Υπάρχουν αρκετά άλλα πράγματα τα οποία ήθελα να πω. Θα σταματήσω όμως εδώ γιατί έχω περάσει κατά ένα λεπτό το χρόνο που μου διαθέσατε. Θα σταματήσω εδώ. Θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις βεβαίως οι οποίες ε, θα προκύψουν και είμαι πολύ ευχαριστώ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς γιατί ήσασταν μέσα στο χρόνο και κατά δεύτερον διότι ήταν απαραίτητο να έχουμε και αυτή την πιο πανεπιστημιακή τεχνική προσέγγιση στο θέμα αυτό, αλλά το κάνατε με πολύ μεγάλη αφοσίωση και νομίζω ότι και εμείς ε, έχουμε ε, κάποια στοιχεία από τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ιγκούε Οφλέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Αφρικανικής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας προσκαλέσατε για να σας παρουσιάσουμε τη θέση μας. Το θέμα του μέλλοντος της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και μετά το 2020 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Αφρική. διότι από τις χώρες μέλη 48, της Αφρικής δηλαδή και Καραϊβικής και Ειρηνικού οι 46 είναι αφρικανικές χώρες. Άρα βαραίνουν πολύ στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Η Αφρικανική Ένωση όμως ε, δεν συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις, ούτε σε επίπεδο και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας του καθεστώτος παρατηρητή που έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως θα γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό εταίρος για την Αφρική. Όμως, η συνεργασία αυτή διέπεται από διάφορα μέσα εταιρική σχέση. Υπάρχει η κοινή στρατηγική Αφρικής Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίθηκε το 2007 στην Πορτογαλία που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική. Υπάρχει συμφωνία Κοτονού, υπάρχει η πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βόρεια Αφρική, υπάρχει και ένα ειδικό μέσο για τη Νότια Αφρική. Συνεπώ, βλέπετε ότι υπάρχει ένα κατακαιρματισμό γεωγραφικό όσον αφορά τις σχέσεις Αφρικής με τον πιο σημαντικό εταίρο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο καθιστά πιο εύθραυστη την διαδικασία ολοκλήρωσης στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν λέω ότι είναι η κύρια αιτία, η μόνη της αργής διαδικασίας ολοκλήρωσης στην Αφρική, αλλά συνεισφέρει στην καθυστέρηση. Αναφερθήκατε σε πολλά σημαντικά ζητήματα και εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας τι κάνει η Αφρικανική Ένωση για τον συντονισμό στην Αφρική. Θα θυμόσαστε ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου ε, Υπουργών το 2006 που εναρμονίζει την κατάσταση και δέχεται 8 κοινότητες περιφερειακές. Υπάρχει μια δικασία αναρμόνισης ε, λοιπόν. Η ΟΚΕ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της Αφρικανικής Ένωσης. Έλεγα λοιπόν ότι ο κατακαιρματισμός αυτός ο γεωγραφικός ε, εμποδίζει την Αφρικανική ολοκλήρωση. Υπάρχουν πολλές παράλληλες διαδικασίες, κάτι το οποίο περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ε, διαφόρων πολιτικών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εταιρική σχέση και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και η Αφρικανική Ένωση ζητάει επίμονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την Αφρική σαν μία οντότητα αδιέρετη στην εταιρική σχέση που έχει. Και αυτό ακριβώς ε, εγκρίθηκε στη Λισαβόνα το 2017. Οπότε ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την βούλησή της αυτή να αντιμετωπίζει σαν μία οντότητα την Αφρικανική Ήπειρο. Η περιφερειακή διάσταση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις σχέσεις της με την Αφρική και τις χώρες ΑΚΕ μετά το 2020 συνεχίζει να βασίζεται στην ε, ήδη υπάρχουσα γεωγραφική δομή και βάζει στην πάντα τις περιφέρειες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε για έναν μηχανισμό για τη Βόρεια Αφρική. Η Αφρική όμως θα χωρίζεται πάντα στην υποσαχάρια Αφρική και στη Βόρεια Αφρική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Αφρικής ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κοινό μέλλον, οπότε δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. για πολλά θέματα πρώτα πλήττεται η Ευρώπη και μετά αφρικανικέ χώρε. Υπάρχει μετανάστευση, υπάρχουν και πολλά άλλα. Πρέπει να δούμε λοιπόν μαζί να είμαστε ισότιμοι εταίροι και να λαμβάνονται οι υπόψη από τους μεν τα συμφέροντα των δε. Η Αφρική προχωράει προς την έγκριση μιας κοινή θέσης για το μέλλον της ομάδας ΑΚΕ. Σήμερα, αύριο στο Κιγκάλι, ξεκινάει μια έκτακτη διάσκεψη των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων των Αφρικανικών χωρών. Και θα ανακοινωθεί εκεί ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στην Αφρική και θα υπάρξει και η έγκριση της τοποθέτησης για το μέλλον των σχέσεων και. Και θέλω να αναφερθώ και να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία της αφρικανικής κοινή θέση. Έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που οδήγησαν σε μεγάλες αλλαγές τόσο στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη. Το πλαίσιο δεν είναι πια αυτό που ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 70. Οι εταίροι επίσης πρέπει να εξελίσσονται, να λάβουν υπόψη τις επιθυμίες και τις ανησυχίες ημέν των ΔΕ. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο λοιπόν για να προωθηθεί μια πιο δίκαια εταιρική σχέση, περισσότερο ισορροπημένη και να μην υπάρχει παραδοσιακή στάση δωρητής δικαιούχος. Εγκρίναμε τους στόχους του 2063, μετά δηλαδή από 50 περίπου χρόνια. Οι στόχοι αυτοί με πολιτικές και προγράμματα στον τομέα της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της ασφάλειας, της διακυβέρνησης, της ανάπτυξης υποδομών κλπ. θα καταστήσουν τη βάση των σχέσεων συνεργασίας της Αφρικής με τους διάφορους εταίρους της. Συνεπώς η Αφρική έχει καθορίσει τις δικές της προτερότητες και μάλιστα σήμερα το απόγευμα φαίνεται εδώ από τα όσα ακούσαμε στο πρώτο πάνελ που ακούσαμε πόσο προχωράει η σχέση Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η Αφρικανική Ένωση αντιμετωπίζεται σαν ένας τρίτος. Θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι υπάρχει άλλη Αφρική στην Αφρικανική Ήπειρο και άλλη Αφρική εδώ στην Ευρώπη από αυτά που ακούμε. Δεν είναι όμως έτσι. Μία είναι η Αφρική. Και οι αποφάσεις αφορούν ολόκληρη την Αφρική. Η κοινή μας θέση είναι η ενότητα της Αφρικής. Η Αφρική πρέπει να μιλάει με μία φωνή. Και ακούσαμε για τη συμφωνία του 2017 που προβλέπει την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο υπήρων που πρέπει να διέπεται από τέτοιες αρχές. Στο Μπιτζάν πριν από τέσσερις μήνες περίπου επιβεβαιώθηκε αυτή η αρχή για να δοθεί νέα όθηση στην εταιρική σχέση. Συνεπώς, η εταιρική σχέση Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινή στρατηγική πρέπει να ενισχυθεί και να αποτελέσει το μοναδικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο υπήρων, Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να συμμετέχουν όλες οι αφρικανικές περιφέρειες και οι πέντε, η Οικονομική και Περιφερειακή Ένωση, αλλά και τα μέλη που αποτελούν την Αφρικανική Ένωση. Και φυσικά να χτίσουμε στα κεκτημένα των διαφόρων μηχανισμών συνεργασίας κοτονού, γυτνίαση κλπ. Άλλη αρχή είναι η πρόθεση της υπηρετικής διάστασης της εταιρική σχέσης. Οι διαπραγματεύσεις τώρα προσφέρουν μια πολύ καλή ευκαιρία για την εξέλιξη αυτή. Σήμερα οι στρατηγικοί εταίροι πρέπει να ασχοληθούν με το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές. Τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που αφορούν την Αφρική και που εξετάζονται εκτός αυτού του πλαισίου. Οι εμπορικέ σχέσεις, για παράδειγμα, ενώ στο Κιγκάλι μιλάμε για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Συνεπώ αυτή η διάσταση η διπυρωτική θα βοηθήσει στην αναρμόνιση των πολιτικών και των δράσεων, θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τη εταιρική σχέση και θα συμφωνήσει ότι έτσι θα υπάρχει και περισσότερη συνοχή στι σχέσει μεταξύ των δύο υπήρων. Πρέπει να προηθηθεί λοιπόν η σχέση αυτή και εμείς επιμένουμε στην αλληλεγγύη μας απέναντι στην περιφέρεια της Καρυβικής και του Ειρηνικού. Και τελώνω λέγοντα ότι η Αφρική είναι μία ήπειρο σήμερα. Είναι προ το συμφέρον όμως και των δύο πλευρών η εταιρική αυτή σχέση. Καλώς σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Μιλήσατε για τον κατακαιρματισμό, για τις ε, σχέσεις χωρών ΑΚΕ Ευρώπης, για την Αφρικανική Ένωση, είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το κατακαιρματισμό και η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής να γίνει πιο επαρκής, πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Jean-Pierre Ελόν Μπασί. Έχετε το λόγο και εσείς 7-8 λεπτά παρακαλώ, ή δυνατόν. Ναι, ή δυνατόν, λέει ο μιλητής. Και εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στην ακρόαση αυτή. Σας χαιρετίζω εκ μέρους του Πρόεδρου μου, του Καλήθου Αμπαπακασάρ Σάλ, δήμαρχο του Ντακάρ, που είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Αρχών της Αφρικής. Η οργάνωσή μας συγκεντρώνει 50 περίπου εθνικές οργανώσεις και 2.000 πόλεις. Και μαζί μέσω των μελών. Είμαστε περίπου 350 εκατομμύρια Αφρικανών πολιτών. Λαμβάνω εδώ το λόγο ως Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης αυτής. Και θέλω να σας πω ότι θα ασχοληθώ με τέσσερα σημεία για να σας εξηγήσω τι μας απασχολεί. Το πρώτο είναι τα μαθήματα που παίρνουμε ως τοπικές αρχές από την εμπειρία που έχουμε από την εφαρμογή της Συμφωνίας του Κοτονού. Το δεύτερο έχει να κάνει με την άνοδο ενό καθεστώτος τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διεθνή σκηνή. Το τρίτο μου σημείο είναι το τι προτείνουμε για μετά το κοτονού. Και το τέταρτο σημείο μου είναι τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μετά το Κοτονού. Όσον αφορά τη συμφωνία της Κοτονού. Για μας, τις τοπικές αρχές, η πιο σημαντική καινοτομία στη σχέση συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ, σε σχέση με τα προϋπάρχοντα, έτσι με τη Συμφωνία Λομέ και η καινοτομία λοιπόν αυτή ήταν η διεύρυνση της αρχής της εταιρική ε, σχέσης για να συμπεριλάβει και άλλους φορείς πέρα από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν πολλά άρθρα που εξηγούν τι είναι αυτή η εταιρική σχέση και γιατί υπάρχει αυτή η διευρυμένη. Γιατί για να υπάρξει ε, να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη ο ρόλος των διαφόρων αυτών εταίρων, να προωθηθεί επίσης η διαδικασία ανάπτυξης και για να βελτιωθεί η καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της στόχιας. Η αρχή αυτή Όμως, συνοδεύτηκε από μεγάλη αμφισημία όσο περνούσε ο καιρός. Τελικά, όλα τα επίπεδα, εκτός από τις τοπικές ε, κυβερνήσεις, θεωρήθηκαν μη κρατικές αρχές. Και αυτή η μη κρατική φορείς στη συνέχεια συμπεριέλαβαν και τις τοπικές αρχές, οι οποίες όμως είναι κρατικές αρχές. Υπήρξαν μηχανισμοί προκειμένου να συμπεριληφθούν, υπήρξαν ε, χρηματοδοτικά μέσα και υπήρξαν ακόμα και θεσμικοί ε, και θεσμικά φόρουμ όπως είναι το ACP Business Forum ή το ACP Civil Society Forum. Οι τοπικές ε, αρχές όμως δεν επωφελήθηκαν από πολιτικό διάλογο ούτε από διαβουλεύσεις στις διαπραγματεύσεις που είχαν να κάνουν με τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα, για παράδειγμα ποτέ επίσης δεν συμμετείχαν στον ορισμό της σχέσης παρά το γεγονός ότι επίμονα το ζήτησαν ξανά και ξανά. Μόνο το 2013, με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφερόταν στην ενίσχυση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για ενισχυμένη διακυβέρνηση και αποτελέσματα αναπτυξιακά πιο σημαντικά, για πρώτη φορά αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι πρόκειται για κρατικούς ε, φορείς, ότι οι τοπικές αρχές δηλαδή είναι κρατικοί φορείς. Και ε, σιγά σιγά δίνεται όλο και περισσότερο χώρος στις τοπικές αρχές. Με τη δική μας την πίεση εγκρίνεται τελικά το 2014 από τους επικεφαλείς ε, κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής η Αφρικανική Χάρτα για τις αρχές της αποκέντρωσης και δημιουργείται και ένα Συμβούλιο των ε, Δήμων και Περιφερειών. Καταλήξαμε σε αφρικανικές θέσεις, επίσης όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους που συζητήθηκαν το 2016 και το 2017, Δημιουργήθηκε επίσης η Global Task Force με την πρωτοβουλία της οργάνωσής μας των ΗΠΑ και τοπικών αρχών, δηλαδή της Αφρικής. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε το στόχο 11 για τις βιώσιμες πόλεις και έχουμε και ό,τι χρειάζεται για να ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας και η μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Για μας λοιπόν, και έρχομαι στο τρίτο, τι είναι το μετά το κοτονού, μετά τη συμφωνία του κοτονού πρέπει να υπάρχει ένα εντελώ διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι είχαμε στη Συμφωνία Κοτονού. Πριν όλα ήταν για την ε, φιλελευθερωποίηση, για την παγκοσμιοποίηση. Σήμερα υπάρχουν πολλέ αμφιβολίες και για τα δύο. Και γι' αυτό πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο του τόνου. Σήμερα οι τοπικέ αρχέ αναγνωρίζονται σαν βασικό παράγοντα τη ε, αλλαγή ε, στην κοινωνία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μα αγνοήσει. Επιθυμούμε λοιπόν, όσον αφορά την Αφρική, τουλάχιστον, στα πλαίσια της ανανέωσης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ μας, πρώτα απ' όλα όντως να αντιμετωπίζετε η Αφρική σαν μία ενιαία οντότητα. Είναι κάτι που στηρίζουμε κι εμείς. Έπειτα, στην αντιμετώπιση αυτή πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές αρχές. Αυτό είναι απέτηση. Και οι τοπικές αρχές πρέπει να εμφανίζονται σε όλες τις πολιτικές και να συμμετέχουν σε όλες τις πολιτικές. Επίσης, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αποτελούν μέρος των χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών μετά το 2020. Για μας χρειάζεται ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός ο οποίο να στηρίζει τη συνεργασία με την Αφρική. Ανησυχούμε όλους ιδιαίτερως για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, γιατί δεν αναγνωρίζεται ο πολύτιμος ρόλος των τοπικών αρχών. Δεν γίνεται μία, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλητής στην ιδέα της επικουρικότητας, εδώ δεν βλέπουμε αρκετά. Πρέπει λοιπόν ο ρόλος των τοπικών αρχών να ενσωματωθεί πλήρως στη Νέα Συμφωνία. Οι τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκές και οι αφρικανικές, έκαναν στην τελευταία διάσκεψη μία πρόταση. Προκειμένου οι τοπικές αρχές να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Έτσι κι τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική η διαδομή υπάρχει και δεν υπάρχει καμία διαφορά, δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε καμία διαφορά. Έφτασε η ώρα, η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δούνε στον αυριανό κόσμο ποιο θα είναι το βάρος τους και συνεπώ πρέπει να έχουν μια συνεργασία, μια ειλικρινή συνεργασία με σεβασμό και αυτή μπορεί να προσφέρει πολλά στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν ε, πάρα πολύ κύριε Ζόμπιε Λομπάζη που δείξατε αυτό το θέμα το πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι στην ε, κοινοβουλευτική συνέλευση ε, μας απασχολεί αυτό και είναι επίσης ε, σημαντικό το ότι το ε, συνδυάσατε με τον υπαριθμό 11 στόχο από τους στόχους της κυλίτιας. Κανονικά οι κυρίες προηγούνται, αλλά τώρα είναι τελευταία η κυρία, η κυρία Κάριν Σοχέτ από την Concord. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την άποψη της Concord, της Ομοσπονδίας ε, των ΜΚΟ. Όποιο και είναι το θεσμικό πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ε, χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι θα είναι μια εταιρική σχέση αρχών ε, ανάμεσα σε ίσους ε, και επίσης το θα λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα, του στόχους και τις πολιτικές προτεραιότητες όλων των εμπλεκομένων. Με αυτά κατά νου Καταρτήσαμε, καταθέσαμε συστάσεις ε, για την ε, εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις αυτές στην ιστοσελίδα μας. Ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπηρετηθούν ε, μακροχρόνιοι στόχοι της ευημερίας, της ειρήνης για όλους ε, και πρώτα απ' όλα να μπουν οι άνθρωποι και ο πλανήτης και μετά να επιδιωχθούν οι στόχοι του θεματολογίου 2030. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι τα θεμέλια θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία και υποχρεώσεις και των δύο πλευρών όπως επίσης και τις συνέπειες ε, της ε, μη συμμόρφωσης. Πρέπει επίσης να υπάρχει σαφής αναφορά στις ε, συμβάσεις των ΗΕ, στο διεθνές δίκαιο και σε άλλες διεθνείς δεσμεύσεις που αφορούν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ε, εξάλλου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, να υπάρχει ιδέουσα προσοχή προς τις πολιτικές τους επιλογές και προς τις αναπτυξιακές τους προτεραιότητες. Όπως επίσης και στην περιφερειακή, στις περιφερειακές πρωτοβουλίες ολοκλήρωσης. Αυτά οφείλουν να ισχύουν για τις τρέχουσες αλλά και για τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στις έξι στρατηγικές προτεραιότητες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, ανθρώπινης ανάπτυξης. Εμείς όμως συστήνουμε να εγκαταλειφθεί η τρέχουσα προσέγγιση ε, και να προκύψει μια άλλη με τρεις ε, διαστάσεις με βάση την αρχή ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπεται να προαχθεί η ευημερία μέσα στα όρια του πλανήτη. Επίσης, θεωρούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι υιοθετούμε τις απόψεις των χωρών και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε πιο ισορροπημένες στόχους και δεσμεύσεις, κυρίως στους τομείς της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων. Ας επανέλθουμε όμως σε αυτή την εταιρική σχέση πολλών εταίρων. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο αλλά και δυνατόν αυτή η συνεργασία να περιλαμβάνει πολλούς ε, παίκτες και ενδιαφερόμενους. Συμφωνούμε από αυτό με τον Ζαν Πιέρ. Υπάρχουν όμως για αυτό τρεις προϋποθέσεις. Η μία είναι να αναγνωριστεί η συνεισφορά του κάθε ε, παράγοντα, ε, να υπάρχει ίση συμμετοχή. Είναι σημαντικό να υπάρχει διαφοροποίηση κυρίως ανάμεσα στο ρόλο των ε, κερδοσκοπικών οργανισμών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ε, και της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών πρέπει να βασίζεται και στους ορισμούς που υπάρχουν για την κοινωνία των πολιτών, ορισμοί των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή αυξάνεται όλο και περισσότερο η κριτική, αυξάνεται και περιορισμοί για τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να οριστεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας έκφρασης, ε, ειρηνικής συνέλευσης και του συνεταιρίζεις αυτά να συμπεριλαμβάνουν και τη δυνατότητα να λαμβάνει κανείς ε, κονδύλια και χρηματοδοτική χρηματική ενίσχυση. Και αυτά να αποτελούν ε, το επίκεντρο των δεσμεύσεων. Όπως είπε και ο Ζαμπιέρ, δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε το ρόλο των ιδιωτικών φορέων όπως ε, αναφέρεται στο άρθρο 4. Η εμπειρία του 2000 δείχνει ότι είναι πολύ εύκολο να χάσει κανείς τις ε, καλές ε, προθέσεις. Ένα βασικό προαπαιτούμενο για ουσιαστική πολυμερή εταιρική σχέση είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, όπως επίσης και το συμφέρον να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών φορέων. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, κυρίως εκεί που προετοιμάζονται τα προγράμματα, ελέγχονται και αξιολογούνται. Εξάλλου όλα αυτά απαιτούν διαφανείς και προσπελάσιμες πληροφορίες, ένα μηχανισμό λογοδοσίας για την εφαρμογή της εταιρικής σχέσης να συνοδεύονται με κοινοβουλευτικό έλεγχο, να μπορεί κανείς να αξιολογήσει πώς ακριβώς λαμβάνονται υπόψη τα απαραίτητα στοιχεία τέτοιοι μηχανισμοί λογοδοσίας πρέπει να περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα για τους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ιδιωτικούς φορείς να καταθέτουν ενστάσεις σε περίπτωση ε, που ε, παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απεραίουν από ε, δεσμευτικές συμφωνίες. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απολύτω απαραίτητα για μια πολυμερή εταιρική σχέση και πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο τη συμφωνία. Αλλά όπω σα είπα ήδη, για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα πρέπει να συνοδεύονται από έναν σταθερό μηχανισμό συμμετοχή σε διάφορα επίπεδα. Αν όλα τα μέρη στη συμφωνία ε, το εννοούν σοβαρά σχετικά με τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, πρέπει να είναι όλοι πρόθυμοι να συμπεριλάβουν και μηχανισμού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και αυτοί, αυτό να το στηρίξουν και με διοικητικά και χρηματοδοτικά μέτρα. Εδώ ε, οι μηχανισμοί που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών περιλαμβάνουν και τέσσερα συμπληρωματικά στοιχεία. Πρώτον, ε, το να υπάρχει συνεισφορά της κοινωνικής της ε, κοινωνίας των πολιτών, στον πολιτικό διάλογο, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεύτερον, η προαγωγή του διαλόγου και των κοινών δράσεων μέσα στην κοινωνία των πολιτών, ανάμεσα στις ε, διάφορες κοινωνίες πολιτών και σε κοινούς ε, κοινοβουλευτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων και των συναντήσεων για να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Τρίτον, όλα αυτά μπορούν να στηριχθούν με ε, online πλατφόρμες για την ανταλλαγή πληροφοριών, για συζητήσεις, για συντονισμό. Και τέλος, να υπάρχουν πιο επίσημοι φορείς κοινωνίας των πολιτών για κάθε περιοχή, έτσι ώστε οι εκπρόσωποι της κοινωνία των πολιτών που θα ορίζονται από τους ομολόγους τους να διατηρήσουν τον κανονικό διάλογο με ανώτερα στελέχη, με υπουργούς και με αρχηγούς κρατών. Οι απόψεις αυτές είναι σε προκατακτική φάση και γι' αυτό θέλουμε αυτά να τα συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας από την κοινωνία των πολιτών των χωρών και, και αργότερα θα επανέλθουμε σε εσά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο πράγματα να υπογραμμίσω. Πρώτα, οι άνθρωποι και ο πλανήτης. Ευχαριστούμε πολύ ε, για αυτό που είπατε και το δεύτερον που είπατε ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Ο ρόλος μας λοιπόν στο Κοινοβούλιο είναι να προστατεύσουμε το χώρο της, ε, των κοινωνιών των πολιτών. Τώρα λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Η πρώτη είναι η Μαρία Χόλμπουργ και θα ακολουθήσουμε η επόμενη. Η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Καμπόνε, Καρμπόνε. Είπατε ότι δεν αυξήθηκε το διαπεριφερειακό εμπόριο. Κατά την άποψή σας, πού οφείλεται αυτό διαπεριφερειακό εμπόριο. Ποια είναι τα αίτια, αυτό με ενδιαφέρει. Οφείλεται ενδεχομένως στο ότι ε, το εμπόριο από αυτές τις χώρες πάει περισσότερο προς την Ευρώπη ή υπάρχουν άλλα αίτια. Ε, κύριε Φλέ, είπατε ότι έχετε την αίσθηση ότι η Αφρικανική κυριε έχει καθεστώς παρατηρητή, η Αφρική είναι κατακαιρματισμένη και για σας ε, το αποτέλεσμα είναι ότι η συνεργασία Αφρικανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Χρειαζόμαστε μία κοινή στρατηγική. Αυτή τη στρατηγική την αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο του κοτονού. Ότι δηλαδή δημιουργούμε κάτι το καινούριο ή μήπως αυτή τη στρατηγική την εντάσσεται σε, αυτό, σε αυτή την ομπρέλα που ανοίγει τώρα ε, έτσι ώστε από κάτω να μπει όλη η ΑΚΕ. Για μας τους πράσινους ανέκαθεν ε, επικρατούσε η άποψη ότι τώρα ε, θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας και εμένα με ενδιαφέρει αν αυτό θέλετε να το ξεκινήσετε από την αρχή ή αν θέλετε να συνεχίσετε με τις χώρες ΑΚΕ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι χώρες ε, ΑΚΕ όσο είναι αυτές δυνατές ως ένωση ε, αποδυναμώνεται η Αφρικανική Ένωση. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Σεσίλ Χιέγκε. Ευχαριστώ πολύ, Νόρβερτ. Να ευχαριστήσω και πάλι τους ε, ομιλητές για τη συνεισφορά τους. η ερώτησή μου είναι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ξέρω καταρχάς να εκφράσω την πικρία μου για την προηγούμενη συζήτηση, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν θα υπάρχει πλέον ε, η κοινοβουλευτική συνέλευση, ε, διότι από ό,τι κατάλαβα θα ακολουθήσουμε τη θεματολογία λίγο. Δηλαδή αυτή η συνέλευση την οποία είχαμε φανταστεί να συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, που κάθε έξι μήνες ε, συναντούμε χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, δεν έχει ακόμα καθορισμένη μορφή. Ε, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε υπό ποια σύνθεση θα γίνεται. Και σε συνέχεια αυτού να πω ότι θα ήθελα να ρωτήσω το εξή ε, τον πρέσβη, για να μπορέσω να κατανοήσω και εάν έχετε φανταστεί το ρόλο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά. Τι ρόλο θα διαδραματίζει στις επόμενες σχέσεις ε, μετά το Κοτονού, διότι αυτή τη στιγμή Υπάρχει μια αντιπροσωπεία Αφρικανικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή θα αντικαταστήσει την ε, συνέλευση. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες επ' αυτού, αλλά να επιστήσω και την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους εδώ στην αίθουσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες ΑΚΕ να πρε... προετοιμαστούν και να αρχίσουν να σκέφτονται προσεκτικά για να μην χωρίσουμε την εξουσία για ένα θέμα το οποίο μας αφορά προσωπικώς. Δεύτερον, Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει θέμα χρόνου και επομένω και χώρου. Δεν ε, ακούω πουθενά να μιλάτε για τη διασπορά στις συζητήσεις. Διότι εμείς έχουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά η διασπορά δεν είναι η κοινωνία των πολιτών. Ο ρόλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου το επιτρέπει, γιατί λέει ότι η διασπορά είναι η έκτη περιφέρεια της Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες χώρες ε, συστήνει μια σειρά από αντιπροσωπείες σε θεσμικό επίπεδο που ε, θα έρθουν να δώσουν φωνή στη διασπορά. Και πρέπει να πούμε ότι η διασπορά από οικονομικής πλευράς έχει πολύ μεγάλη εξουσία, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Εγώ αναφέρθηκα μόνο στον οικονομικό τομέα και θα ήθελα να γνωρίζω ποιος θα είναι ο ρόλος της διασποράς στη συνέχεια μετά το κοτονού. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ακόμα εκκρεμεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η συνέλευση αυτή. Ε, αν την εγκαταλείψουμε θα είναι ολέθριο σφάλμα. Η ισομερή συνέλευση θα είναι εις βάρος της ανάπτυξης της Αφρικής και θα την καταδικάσουμε στην αποτυχία, διότι δεν υπάρχει επιστροφή της πραγματικότητας, ε, θα βρεθούμε ε, με μια συχνά λανθασμένη αντίληψη, το λέω και το επαναλαμβάνω, της ανάπτυξης. Ε, το να πάμε πέραν της συμφωνίας του Κοτονού, κανονικά θα πρέπει να βρούμε τη συμφωνία του Λομέ. Η συμφωνία Λομέ ε, ήταν αυτές οι προνομιακές συμφωνίες εμπορίου και ανάπτυξης που δεν αφορούν μόνο την αγορά, διότι σήμερα έχουμε μια αποτυχία του συστήματος ανάπτυξης και αυτό ε, σε μεγάλο βαθμό ε, οφείλεται σε αυτή την προσέγγιση η οποία ε, ασχολείται μόνο με την αγορά και δεν λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες της ανάπτυξης είτε είναι αποκεντρωμένη είτε είναι κρατική. Είτε γίνεται στα Εμμυράτα, είτε γίνεται στην Ιαπωνία, είτε από εμά προπολεμικά. Ε, τα πάντα γίνονται λόγω της ανάπτυξης και μέσω των κρατών. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε προνόμια σε αυτή την τεράστια πρόκληση, πρέπει να βρούμε την οδό και τα μέσα για μια κοινή ανάπτυξη. Εγώ που εργάζομαι σε ιδιωτικό επίπεδο ε, πέραν της εργασίας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει ένα ταμείο για να βοηθήσουν την Αφρική και να εμπλέξουμε και τους ιδιωτικούς παράγοντες, διότι ε, μας ζητούν συνέχεια περισσότερη βοήθεια. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν το κράτος είναι θεμελιώδης σημασία και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Δεν θα υπάρχει ανάπτυξη χωρίς πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και οικονομικό επίπεδο σημαίνει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, στρατηγικό όρομα και όχι βραχυπρόθεσμο όραμα των αγορών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, περάσουμε στα μέλη του πάνελ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μας πει δύο λόγια αν θέλει. Όχι. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Γενική Διεύθυνση Ντεύκο αν θέλει να λάβει το λόγο. Ούτε και αυτή επιθυμεί. Ωραία. Πρέπει να τελειώσουμε το αργότερο στις 5 και 4. Τρία-τέσσερα λεπτά ο καθένα λοιπόν για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και για να ολοκληρώσετε και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, με τον κύριο Καρμπόνε. Ναι, θα ξεκινήσω προσπαθώντας ε, να προκαλέσω και το φίλο μου εδώ από την Αφρικανική Ένωση. Διάβασα την ομιλία του Μουσαφάκη που έκανε χθες και νομίζω ότι είπα αυτά που είπατε κι εσείς. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Εάν αυτή είναι μια νομική συμφωνία, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ότι θα έχει πρόσβαση, θα προσχωρήσει η Αφρικανική Ένωση σε αυτή τη συνθήκη. Και υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα, ρήτρα Ρέγιο, που είναι όμως ε, ε, ε, μία ρήτρα που αφορά έναν περιφερειακό οργανισμό ολοκλήρωσης ε, και έχει το εξής πρόβλημα. Μόνο τα μέλη αυτής της συγκεκριμένη περιφέρειας, αυτής της συγκεκριμένη περιοχής αποφασίσουν να εκχωρήσουν εξουσία σε αυτό το διεθνή οργανισμό μπορεί να ισχύσει. Επομένως μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται την προσχώρηση της Αφρικανικής Ένωσης σε αυτή τη συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά θα περιοριστώ σε αυτό. Και το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι η σχέση μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και των Περιφερειακών ε, Συμβουλίων δεν είναι τόσο ρευστή όσο θέλετε να πιστέψουμε. Συγγνώμη που το θέτω έτσι τόσο ομά, αλλά ε, υπάρχουν συνεχείς εντάσεις μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και των Περιφερειακών Οργανώσεων. Δεύτερον, Είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να διαγράψουμε πλήρως τις χώρες ΑΚΕ. Πράγματι υπάρχει αυτή η ιδέα ότι η νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, φαίνεται ότι δεν έχει κοινή ταυτότητα, κοινή ιστορία, αλλά υπάρχει μόνο κοινό συμφέρον μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Και ένα δεύτερο Είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν άλλα κοινά στοιχεία μεταξύ αφρικανικών χωρών και κάποιων χωρών Καραϊβικής και Ειρηνικού. Τρίτον, είμαστε βέβαιοι ότι ε, ίσως η Αφρική να μην χρειάζεται την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσει στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής, ε, ε Αφρικής, Καραϊβική και Ειρηνικού και να μεσολαβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να απαντήσω και την ερώτηση της κυρίας Χόιμπουχ. Είναι μία από τις σαφείς δηλώσεις που κάνω προς τους φοιτητέ μου και έχω και έναν εδώ στην αίθουσα και τους ρωτάω την ίδια ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότεροι φραγμοί μεταξύ Λιβερίας και Γκάνας ή Λιβερίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση είναι μεταξύ Λιβερίας και Γκάνας. Το, ο λόγος για τον οποίο το ενδοπεριφερειακό εμπόριο είναι τόσο περιορισμένο είναι γιατί υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και οι χώρες ανήκουν σε περισσότερες από μια περιφερειακές οργανώσεις και αυτό δημιουργεί το εξή πρόβλημα, το πρόβλημα της διαφοροποίησης. Οι περισσότερες από τις χώρες που είναι γειτονικές, η μία δίπλα στην άλλη, παράγουν τα ίδια αγαθά και μετά κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω προς την κυρία Κιέγκε και να τα πω ιταλικά, άρα τέλος πάντων να τα πω αγγλικά. Είστε έτοιμοι να ταξιδεύετε τρεις φορές το χρόνο στην Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Γιατί είμαι βέβαιος, με τον τρόπο τουλάχιστον που διάβασα εγώ την ε, ε, πρόταση, ε, τη, συνέλευση, την Έχουμε πιο συγκεκριμένε προτάσεις και συγκεκριμένε συνελευσει μεταξύ κοινοβουλίων. Είστε διατεθειμένοι λοιπόν να ταξιδεύετε σε τρεις διαφορετικούς προορισμούς για να γίνονται συνεδριάσεις των συνελεύσεων, να έχουμε περιφερειακές κοινοβουλευτικέ συνελεύσει. Ευχαριστώ, αλλά μόνο μια φορά το χρόνο ταξιδεύουμε. Να δώσω τώρα το λόγο στο Μοχάμετ Γκουέι οφλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να πω τα ίδια με τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης. Πάντως, να ξέρετε ότι αυτή είναι η θέση μας, η θέση της Αφρικανικής Ένωσης και βέβαια άπαξ και έχει ψηφιστεί, εννοείται ότι θα την μοιραστούμε μαζί σας και με όλους μας τους εταίρους. Πρώτα απ' όλα, και κάτι που είπε ο κύριος Καρμπόνε, δεν υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στην Περιφερειακή Οικονομική Πετροπή και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, η Αφρικανική Αρχιτεκτονική για την Ασφάλεια. Ο καθένας παίζει το ρόλο του. Συγκεκριμένα, Υπάρχει σήμερα μια κρίση στην Αφρική, μια σύγκρουση. Η πρώτη απάντηση είναι η Αφρικανική Ένωση. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 80 με τον ΟΙΕ, παργούς και τα... είναι Αφρικανική απάντηση. Στο Μαλί, στην Κεντρική Αφρική κλπ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Όσον αφορά τις ανταλλαγές, γιατί για το άλλο μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αργότερα αν θέλετε. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές αιτίε. Σήμερα αποφασίζουμε για την ε, υπηρετική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Και σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν από τον ΟΙΕ, αυτή η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για την Αφρική θα έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι το 2022 να διπλασιαστεί ο όγκος. Κάτι το οποίο δίνει λύση και στο πρόβλημα που είχαμε για τον συντονισμό των περιφερειακών οργανώσεων. Πριν υπήρξε μια πληθώρα. Τώρα αναγνωρίζονται 8. Και έτσι υπάρχει και τριμερές, το τριμερές Σαντέκ, ε, Ανατολική Αφρική κλπ. Συνεπώς έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει αυτή η ελεύθερη ζώνη και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τελωνιακή ένωση και η κυκλοφορία ατόμων στην Ανατολική Αφρική είχε γίνει πραγματικότητα. Τώρα δεν έχω χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες. Η κυρία Έρμπες ρώτησε για τον κατακαιρματισμό της Αφρικής. Είναι γεγονός. Δεν είπα ότι θα υπάρξει μια κοινή στρατηγική. Από το 2007 έχει εγκριθεί στη Λισαβόνα. Υπάρχει δεν είπα τίποτα για την αντικατάσταση της Συμφωνίας Κοτονού. Η θέση όμως θα είναι κοινή μεταξύ όλων των εταίρων. Θα γίνει αυτό υπό την αιγίδα και η Αφρική πιστεύει το πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο είναι να υπάρχει εταιρική σχέση μέσω της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από ε, μικτές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Τώρα για να απαντήσω στην κυρία Κέγκερ. Κατά πόσο το Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο θα αντικαταστήσει την εταιρική σχέση πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Η διασπαρόντος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και οικονομικά. Εννοείται. Η Αφρικανική Ένωση έχει καθεδρήσει διάφορες πολιτικές για να ενισχύσει το ρόλο της διασποράς. Τέλος. Για να απαντήσω στον κύριο Σαφοζέ. Και συγγνώμη αν σφαγιάζω το όνομά σας. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμες πολιτικές και όχι βραχυπρόθεσμες. Ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά, ο κύριος Μπάση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να κοιτάμε τα πράγματα κατάματα. Η εφαρμογή της Συμφωνίας Κοτονού οδήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες ΑΚΕ από κοινού κατέληξαν ότι χρειάζεται αυτή η στρατηγική κοινή, γιατί διαπίστωσαν αδυναμίες στον πολιτικό διάλογο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και να αναγνωρίσουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα πιο αποτελεσματικά σύνολα είναι τα υπηρετικά. Ωραία, οι χώρε ΑΚΕ έχουν μια παλιά ιστορία, σύμφωνη, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον ΟΗΕ όταν συζητούμε, συζητούμε με την Αφρικανική ομάδα, με την Καρεβική ομάδα, με την ομάδα Ειρηνικού κλπ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στον ΟΗΕ έτσι γίνεται η συζήτηση. Δεύτερον, σε θέμα τοπικών αρχών. Ο δυναμισμός αυτός ο τοπικός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μέσα στην πραγματικότητα τοπικές αρχές. Κύριε Σοφαζέρ, μιλήσατε για συνανάπτυξη. Όρος που είχε εξαφανιστεί από την ευρωπαϊκή ρητορική τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε στο Λομέ και στη Γιαουντέ. Έχετε το θάρρος να επιστρέψετε, γιατί ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Η Ευρώπη έχει το θάρρος να στηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο και τη διεθνή αλληλεγγύη. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το πρόβλημα αυτό προς το παρόν ε, δεν έχει απάντηση, ενώ αυτή θα έπρεπε να υπάρχει στη νέα συμφωνία. Και θα φροντίσουμε γι' αυτό. Ενθαρρύνουμε τους πρέσβησα και την Αφρικανική Ένωση να υπάρξει μια πραγματική συνανάπτυξη, από κοινού ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπογραμμίσατε τη σημασία της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο και ε, θα ακούσουμε τώρα την άποψη της ε, κοινωνίας των πολιτών. Θέλω να πω κάτι για την κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση, γιατί πράγματι πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας και εμείς ως κοινωνία των πολιτών ε, συνεργαστήκαμε πολύ με την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση, την κοινή. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο μέλλον σε όλα τα επίπεδα, στο περιφερειακό και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Εμείς θέλουμε να έχουμε πολύ καλό ε, διάλογο με τα κοινοβούλια σε όλα τα επίπεδα. Απλά να πω ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία των πολιτών να υπάρχει ένας χώρος περιφερειακός ε, που να έχει προσαρμοστεί στην ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και νομίζω ότι οι εταίροι μας, οι ΑΚΕ, επιθυμούν να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και γι' αυτό πρέπει να ακούμε κιόλα. και γι' αυτό είπα ότι θέλω ε, να ακούσω το τι έχουν να μας πούν τι πιστεύουν για αυτή τη συνεργασία σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Δεν ήταν εύκολο, ε, συστήθηκε ένα φόρουμ ε, κοινωνίας των πολιτών, αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο το να καταστήσει κανείς αυτό το φόρουμ λειτουργικό. Δεν είναι εύκολο αν δεν υπάρχει καμία οικονομική υποστήριξη. Δεν είναι εύκολο να ε, λειτουργεί κανείς σε αυτές τις ε, τρεις μεγάλες περιοχές. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον και δεν πρέπει τόσο εύκολα ε, να το απορρίπτουμε σε επίπεδο χωρώνα και, και, και επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες Νομίζω ότι ακούσαμε διάφορες απόψεις, είναι όλες για μας πολύ χρήσιμες ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο ψήφισμά μας ε, που θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας την επόμενη σάντησή μας στις 24 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας εύχομαι καλό απόγευμα.

Excuse me, maybe we can start with our agenda, because we have couple... Να ξεκινήσουμε για την ημερήσια διάταξη, γιατί έχουμε ένα-δυο σημεία ακόμα. Σημείο 15, Μηχανισμό πολιτική Προστασία τη Ένωση, Μετά έχουμε το μέλλον των τροφίμων και τη γεωργία. Δεν έχουμε και πολλού συναδέλφου εδώ, αλλά τέλο πάντων να ξεκινήσουμε με το 15. Μηχανισμό πολιτική Προστασία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να ενισχύσει την ε, ε, συνεργασία και να έχουμε ευέλικτες διαδικασίες, αλλά η πιο σημαντική αλλαγή είναι να ενισχύσουμε τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστροφές, δημιουργώντας ένα αποθεματικό δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σημαίνει ότι αν εγκριθεί η πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της ε, βοήθεια, για παράδειγμα ε, σχέδια πυρόσβεσης, ε, για να αντιποκρίνονται σε φυσικές καταστροφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν είναι διαθέσιμη εθνική πόροι γιατί αντιμετωπίζουν ε, κρίση. Είδαμε το καλοκαίρι την τεράστια ζημιά που προκάλεσαν οι πυρκαγιές και τη βοήθεια που παρασχέθηκε από άλλα κράτη-μέλη. Ε, και η πρόταση αυτή προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα που υπήρχε. Η πρόταση για μας είναι πολύ σημαντική γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και για κρίση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως φυσικές καταστροφές αλλά όχι μόνον και ε, συνεργάζεται παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, επομένως η σχέση με τα δύο μέσα θα πρέπει να καθοριστεί σαφέστατα. Αρμόδια επιτροπή είναι η ΕΜΒΗ, η συγγήτρια είναι η κυρία Ελίζαμπέτα Γκαρντίνη από το ΕΛΚ και η ΔΕΒΕ είναι συνδεδεμένη βάσει του άρθρο 54. Από την επικροτροπή μας η συντάκτρια είναι η κυρία Ζόφκο και θα μιλήσω εξ ονόματος της κυρία Ζόφκο διότι ζητά συγγνώμη αλλά δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα μαζί μας ε, λόγω υποχρεώσεων που έχει ως επικεφαλής της παρατήρησης, αποστολής αποτήρησης ε, εκλογών ε, στο Νεπάλ που δίνει και συμβουλές στην ε, κυβέρνηση του Νεπάλ. Μας ε, λέει ότι επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ότι παρουσιάστηκε μια πολύ καλά μελετημένη πρόταση για να βελτιώσει τη δυνατότητα ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε καταστροφές, να ενισχύσει και προληπτικά μέτρα τα οποία θα συνάδουν και με άλλα μέσα χρηματοδότησης και θα έχουμε μια απλοποιημένη διαδικασία για την ενεργοποίηση του μηχανισμού. Η γνωμοδότησή της προσπαθεί να ενισχύσει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής ε, ε, πολιτικής και αναπτυξιακής πολιτικής ε, τη σχέση με ανθρωπιστικούς οργανισμούς και με χώρες τρίτες εταίρους για να έχουμε σημαντική συμβολή στο πλαίσιο για τη μείωση των κινδύνων. Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική πτυχή αυτού του μέσου, τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας Πρέπει να γίνεται σαφή διάκριση μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων, ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνοχή μεταξύ διαφορετικών μέσων ως τελικό αποτέλεσμα ε, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση των ε, καταστροφών από ε, φυσικές καταστροφές. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο, διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων και πού υπάρχουν επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας για να μπορέσουμε να έχουμε και θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ουδέτερος παράγων προτείνεται στήριξη της Ένωσης μέχρι το 55% για κόστος μεταφοράς για κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πουλ ε, μέσων ενώ οι δυνατότητες διάσωσης θα είναι υπό την εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξή τους. Ε, επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος ε, της ενίσχυσης των εθνικών μηχανισμών, αλλά θα πρέπει να είναι για κατεπίγουσα δράση, για καταστροφές ε, στις οποίες ε, διαπιστώνουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και να δώσω τώρα το λόγο στη σκιώδη συγγήτρια την κυρία Κιέγγε που είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε που νομίζω ότι θα πρέπει να μας ε, καθοδηγήσουν ε, στο να δώσουμε κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά λοιπόν κάποια θέματα, ε, θα ήθελα να ξεκινήσω από την ε, εμπειρία της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια ήρθε αντιμέτωπη με μία σειρά φυσικών καταστροφών, ξεκινώντας με το σεισμό, αλλά και οι πυρκαγιές, οι οποίες αφορούσαν ε, περισσότερο άλλες χώρες, αλλά σε κάποιο βαθμό και την Ιταλία. Επίσης ε, υπάρχουν και οι υπερχιλήσεις των ποταμών, φυσικές καταστροφές ε, και η Ιταλία μπόρεσε να καταφύγει σε αυτό το μηχανισμό της ε, πολιτικής προστασίας. Επίσης θεωρώ ότι υπήρξαν και κάποιοι άλλοι μηχανισμοί επιτόπου, θα μπορούσαν βέβαια να υπάρχουν ε, κάποιες άλλες υποδομές ε, που θα ε, χρησιμεύουν όχι μόνο για την εκ των υστέρων βοήθεια, αλλά εκ των προτέρων, προετοιμασία, πρόληψη, πώς μπορεί να προετοιμαστεί το, η, χώρα για να υπάρχει ασφάλεια σε περίπτωση υπερχειλήσεων παραδείγματος και πλημμυρών. Και σε αυτό λοιπόν τον τομέα Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συμμετοχή από πλευράς μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Ένα άλλο θέμα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξίσου σημαντικό, είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτή η πρόταση που ετέθη ε, σχετικά με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει αρκετά ουδέτερη όσον αφορά τη διαχείριση δαπανών, όπως είναι οι μεταφορές, το μεταφορικό κόστος. Αυτό θα μπορούσε να καταλογιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα έπρεπε επίση να γνωρίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, να έχει νομοθεσία που να αφορά σε πρόληψη καταστροφών. Ε, εθνική νομοθεσία η οποία τα αφορά στην πρόληψη καταστροφών αλλά να προβλέπει η εθνική νομοθεσία και την παρέμβαση του κράτους. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνω μεταρρυθμίσεις, νομοθεσία, ε, το να εκμεταλλευτεί κανείς τις ε, καλές πρακτικές ε, άλλων κρατών, Ιταλίας αλλά και άλλων. Όλα αυτά να συγκεντρωθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο καλύτερα να μεταρρυθμίσουμε αυτό το σύστημα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω με αυτήν την ε, εμπειρία να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά γιατί αυτό θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό για να βοηθήσουμε τις χώρες εκείνες ε, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ευάλωτες, ε, είναι εγκατρελειμμένες, μόνες τους καλούνται να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι σκιώδεις Γι' αυτό δίνω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστώ και την σκιώδη συγκήτρια. Λίγα λόγια επιτρέψτε μου να πω εν είδη αντίδραση σε αυτά που ελέγχθησαν. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, βεβαίως ε, υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπέγραψε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα σαφές για το ρόλο της πολιτικής προστασίας. Παραμένουμε ε, στους ε, κανόνες που προβλέπει αυτή η συμφωνία. Όσον αφορά την ε, ουδετερότητα, οι περισσότερες εκ των παρεμβάσεών μας αφορούν θεομηνίες, ξαφνικές θεομηνίες, ζώνες εκτός συγκρούσεων. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, επίσης γνωρίζουμε τη σημασία της ε, ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων. Αυτό που δεν βλέπετε ε, από τη φύση του είναι το ότι σε κάποια επίσημα αιτήματα αρνούμεθα γιατί θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία και ουδετερότητα δεν θα διατηρηθούν. Κυρίως όταν παίρνουμε κάποια αιτήματα από διεθνείς οργανισμούς να βοηθήσουμε σε θέματα επιμελητίας, σε εμπόλεμες περιοχές. Για μας ο διαχωρισμός είναι απόλυτα σαφής. Όμως η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία πλέον δεν ε, συμβαδίζουν σε πάρα πολλούς ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσει, απλά αλληλοσυμπληρώνονται. Παραδείγματο χάρη, οι τυφώνες Ήρμα και Μαρία πέρυσι το καλοκαίρι, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ε, συγχρηματοδότησε ένα ε, σκάφος για να μεταφέρει τρόφιμα και άλλο υλικό από ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις, WFP και άλλες. Αυτό εννοώ με συμπληρωματικότητα. Άλλο, άλλο παράδειγμα, στους καταπλησμούς των Ροχίνγκα στο Μπαγκλαντές, κάποιες σκανδιναβικές ή βόρειες χώρες στην ε, Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Εταιρική Σχέση έστειλαν ε, πολύ γρήγορα κοντέινερ στο Κόξ Μπαζάρ. Ε, εμείς ε, συγχρηματοδοτήσαμε ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας και τελικά σε ένα από αυτά τα κοντέινερ υπάρχει και μία ε, σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι δουλεύουμε συμπληρωματικά με τους εταίρους μας και στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ η πολιτική προστασία και το ανθρωπιστικό στοιχείο αφορούν τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση θεομηνιών. Αυτά όμως ε, σε μας είναι συντονισμένα ε, σε ένα και μόνο κέντρο. Για να απαντήσω στην αξιότιμη Ευρωβουλευτή από την Ιταλία, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξής. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που αφορούν, αφορούν στην προετοιμασία του νομικού κειμένου που προτείνουμε. Επειδή όμως η ε, πολιτική προστασία είναι μόνο ο μηχανισμός στήριξης, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, να έχουμε μια συνοδευτική δήλωση όπου να φέρουμε με σαφήνεια ότι η πρόθεσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που προέρχονται από διαρθρωτικά ταμεία και επενδύσεις από διαρθρωτικά ταμεία να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους το θέμα της ε, πρόληψης και της ε, ετοιμότητας. Συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο για να ε, εξελίξουμε περαιτέρω τα προαπαιτούμενα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις έχουν αποτέλεσμα. Ε, πρόληψη, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ετοιμότητα, αυτά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οποτεδήποτε εκταμιεύονται κονδύλια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλετε κάτι να πείτε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την απάντηση που μου εδότη, αλλά θέλω να πω και το εξή. Σε πάρα πολλέ από τι περιπτώσει που αναφέρθηκαν, νομίζω ότι η Ιταλία κατέφυγε ε, στο αποκαλούμενο Ταμείο τη Αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν μα βοήθησε να ξεφύγουμε. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή όπου πριν από 6 χρόνια είχαμε το σεισμό και αν πάτε τώρα σήμερα, αν δείτε όλα αυτά τα έργα που έχουν λάβει χώρα, έργα οικοδόμησης. αυτά έλαβαν χώρα ακριβώς με κονδύλια του Ταμείου Αλληλεγγύης. Άρα δηλαδή μπορούμε να συνδυάσουμε ε, τα διευθυντικά ταμεία με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αυτό το κάναμε εμείς ε, και υπήρξαν ε, πολλές παρεμβάσεις, όποτε, οποτεδήποτε είχαμε φεμινίες και στη δική μου την περιοχή, αλλά και στον τελευταίο σεισμό. Υπήρξε λοιπόν συνδυασμός αυτών των κονδυλίων και γι' αυτό σας ευχαριστώ και για την απάντησή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Και στην εισηγήτρια θα στείλω όλα αυτά τα μηνύματά σας και τις λύσεις που προτείνετε. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 22 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν. Πρόκειται για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Η συγγήτριά μας μόλις έφτασε. Συντάκτρια γνωμοδότησης. Οπότε θα σας δώσω και το λόγο. κύριε Νόικλου. Αρμόδια επί της ουσίας είναι Επιτροπή Γεωργίας για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Με τον Herbert Orphan από το η 29 Νοεμβρίου η Επιτροπή πρότεινε διάφορα μέτρα με ανακοίνωσή της που προτείνουν αλλαγές για την ΚΑΠ προκειμένου αυτή να απλοποιηθεί και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε πιο καλά αποτελέσματα. Στα τέλη του Μαΐου του 2018 θα πρέπει να έχει εγκριθεί. Γι' αυτό και εμείς θα ψηφίσουμε στις 16 Μαΐου του 2018 προκειμένου να καθορίσουμε την κατεύθυνση της νέας ΚΑΠ. Λοιπόν, συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η κυρία Νόικλ από τη δικιά μας την Επιτροπή. Σας ακούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να πω μόνο λίγα λόγια. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική αντιμετωπίζεται πολύ συχνά ως μια πολιτική που αναφορά μόνο την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια, ούτε και έτσι εμείς ε, εννοούμε την γεωργική πολιτική, ε, το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε. Αυτό έχει επιπτώσει στις χώρες του Νότου, κυρίως ε, σε χώρες στις οποίες μεταφέρουμε προϊόντα ή παίρνουμε προϊόντα από αυτές. Άρα δηλαδή υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα ε, στις πολιτικές αυτές. Δεν θα αναφερθώ σε καταναλωτικές συνθήκες, αλλά περισσότερο στις επιπτώσεις ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν στην έκθεσή μου αναφέρω ότι χρειαζόμαστε μια συνεπή πολιτική, γιατί δεν είναι δυνατόν η γεωργική ή η αλλιευτική πολιτική να στρέφονται κατά των αναπτυξιωμένων χωρών και μετά εκ των υστέρων να προσπαθούμε να τα μπαλώσουμε με την αναπτυξιακή πολιτική. Σημασία έχει να αισθανόμαστε δεσμευμένοι ως προς τους στόχους της χιλικής, κυρίως με τον στόχο υπαριθμών 2 που αφορά την πείνα ή τον στόχο υπαριθμών 12 καταναλωτικές συμπεριφορές συμπεριφορές ή ε, στόχος 15, ζωή στην Ήπετρο. Αυτοί οι στόχοι πρέπει απαρέγκλιτα να στηριχθούν και πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι κατά κάποιο τρόπο εξαρτώνται από τη δική μας γεωργική πολιτική. Στα σημεία 3 και 4 αναφέρω ότι υπάρχουν χώρες από τις οποίες εισάγουμε προϊόντα, μεταξύ αυτών η Βραζιλία. Σε μεγάλο βαθμό εισάγουμε σόγια. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι και το σωστό. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν είναι σωστό. Μακροπρόθεσμα ε, πρέπει να καλλιεργούμε τις δικές μας εκτάσεις, ε, να μην ε, κάνουμε κατάχρηση και να μην ε, εισάγουμε σόγια από αυτές τις χώρες. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εντάξει αυτό είναι καλό για τις χώρες ότι κάνουν εξεγωγές. Όμως όλοι που είμαστε εδώ γνωρίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό προκύπτει εσωτερικός εκτοπισμός ε, πληθυσμών, χάνονται θέσεις απασχόλησης, εξαφανίζονται οι μικροί γεωργοί. Άρα δηλαδή όταν αγοράζουμε σόγια ας πούμε από μια χώρα, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό για το σύνολο των πολιτών, ίσως για λίγους. Το ίδιο, το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές μας, ε, γιατί εξάγουμε ε, πουλερικά και ντομάτες, παραδείγματος χάρη, σε αδύναμες αγορές. Εξαγωγές σε αδύναμες αδύναμες αγορές σημαίνει ότι αυτές οι αγορές δεν θα ενισχυθούν στο μέλλον. Έχουμε αίμα στα χέρια μας και να το πούμε αυτό. Παραδείγματο χάρη ε, το γάλα της Βαβαρίας, τι δουλειά έχει στην Μπουρκίνα Φάσο. Να βοηθήσουμε καλύτερα τους καλλιεργητές στην Μπουρκίνα Φάσο μόνοι τους να καλλιεργούν τα προϊόντα τους, όχι να τους ε, πουλάμε τα δικά μας. Πολλοί λένε ότι ε, κύριε Χόγκεν, ε, ας πούμε, ο Επίτροπος, ότι πρέπει να επεκτείνουμε τις αγορές μας. Εσείς είστε Επίτροπος Γεωργίας, κύριε Χόγκεν, και η δουλειά σας είναι όχι μόνο να αυξάνετε τις εξαγωγές, αλλά ε, να έχουμε μια καλύτερη δική μας ε, βιώσιμη γεωργία πρέπει να τονίσουμε ότι ο μύθος αυτός, το αφήγημα ότι η Ευρώπη οφείλει να θρέφει τον υπόλοιπο κόσμο, αυτό πρέπει να πάψει. Ε, λένε ότι να αυξήσουμε την παραγωγή μας ε, για να χορτάσουν όλοι. Λάθος αυτό. Εμείς ε, δεν έχουμε πρόβλημα ποσοτήτων, έχουμε πρόβλημα κατανομής. Τέλος λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι εμείς οφείλουμε να θρέψουμε όλο τον κόσμο. Και επίσης καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τους στόχους της χιλιετίας να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων, να διαπιστώσει ότι και η ΓΚΑΠ, η κοινή γεωρική πολιτική φταίει. Η κοινή γεωρική πολιτική φταίει και αυτή για την πείνα στον κόσμο. Φταίει που έχουμε μεγαλύτερη μετανάστευση, ως εκ τούτου στην Ευρώπη πρέπει να βρούμε μια τέτοια γεωργική πολιτική που θα καθιστά τους γεωργούς υπεύθυνου να αναλαμβάνουν, και αυτοί τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Οι σκιώδεις τώρα. ΕΛΚ. Εγώ θα μιλήσω εκ μέρους του κύριου Κώσσα, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Όμως, θέλει ο κύριος Κώσσα να ευχαριστήσει την συντάκτρια της γνωμοδότησης. Υπάρχουν κάποια σημεία στη γνωμοδότηση αυτή που είναι προβληματικά για την ομάδα του ΕΛΚ. Το σημείο 3, για παράδειγμα, που ζητά ένα νέο κεφάλαιο στην ε, κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 που εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Σημείο 5. Ζητάει αλλαγή αντί να γίνονται οι ενισχύσεις ανά έκταση, πρέπει να συνεχίσουμε όπως τώρα, γιατί εξαιτία της φύση τους ενισχύσεις αυτές είναι βολικές και εφαρμόζονται και πιο εύκολα. Και στο σημείο 6, ο Σκιώδης εισηγητής, δεν πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει την ευθύνη για, την, ε, ε, για να ταΐσει μάλλον τον ε, κόσμο. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γεωργική πολιτική που να βοηθάει την ανάπτυξη της Ευρώπης. Πρέπει να διασφαλίζει η ικανή παραγωγή τροφίμων, να υπάρχει βιώσιμη διαχείριση των πόρων και της κλιματικής δράσης και να συνεισφέρει σε μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Γι' αυτό και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη νέα γνώση, νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα. Και αυτό δεν είναι μύθος, είναι το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ. Τώρα οι άλλοι σκιώδεις. Η Μαρία πρώτα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να στηρίξω ανεπιφύλακτα τη Μαρία Νόιχελ. Τέλειωσες λέγοντας ε, ότι ε, να αναλάβουμε την ευθύνη και την ευθύνη για τους ε, γεωργούς της αναπτυσσόμενης χώρες, όχι μόνο για τους δικούς μας. Και εγώ όμως θέλω από αυτού να πω ότι εμείς ευθύνη να αναλαμβάνουμε ούτε για τους δικούς μας γεωργούς, ούτε για τους άλλους. Ε, κάθε μέρα χάνουμε στην Ευρώπη εκατοντάδες ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είμαστε μέσα σε μια περιδίνηση όπου κατ' ουσίαν οι γεωργοί τρέχουν πίσω από την ανάπτυξη. Εισαγωγές λοιπόν και εκεί συμφωνώ μαζί σου, εισάγουμε πρώτες ύλε κατά κύριον λόγο και μετά εξάγουμε μεταποιημένα προϊόντα. Και κάπου στη μέση βρίσκονται οι μεσάζοντες, ε, αυτοί δεν είναι οι ούτε και στον Νότο. Σε μια τέτοια γνωμοδότηση, επειδή δεν υπάρχει περιθώριο ε, στην έκταση της γνωμοδότησης, μπορούμε να επισημάνουμε αρκετά θέματα για να είμαστε πιο αυστηροί. Ε, στο είπα και πριν, συμφωνώ μαζί σου, ε, τα είπες αυτά που σκέφτομαι και εγώ. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες, όχι με τη μορφή κριτικής, αλλά για να γίνει η γνωμοδότηση πιο ισχυρή. Να πω το εξής, όσον αφορά αυτά που είπε ο εισηγητής εισηγητής, και ο εισηγητής ε, από το ΕΛΚ. Ξέρετε κάτι, εχθές ε, στην ε, Επιτροπή Ελέγχου των Προεπολογισμών είχαμε συζήτηση σχετικά με τις γεωργικές ενισχύσεις, το πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να κάνουμε εξοικονομίες αυτό που έχει ενδιαφέρον, ακριβώς ε, οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ είπαν ότι στις ενισχύσεις δαπανάμε χρήματα γιατί κάνουμε πλούσιους ε, τους ε, πιο, τους πιο πλούσιους. θεωρώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει κάπως να αλλάξει και ειδικά όσον αφορά αυτό σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο, αν αναλάβουμε την ευθύνη για πολιτικά θέματα, τότε θα ε, επιτύχουμε τους στόχους της χιλιτίας και θα βοηθήσουμε και τους ε, γεωργούς τόσο εδώ όσο και στο νότο σε ολόκληρο τον κόσμο. Μαρία, χαίρομαι που συνεργαζόμαστε και στο τέλος θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλετε το λόγο, όχι. Εντάξει, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε. Ο κύριος Κλάρκ από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξη σήμερα. Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική κάθε άλλο παρά τέλεια είναι και θα προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο στην επόμενη μεταρρύθμιση. Να είναι πιο βιώσιμη, να είναι πιο αναπτυξιακή και να εφαρμόζει και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, επίσης μπορεί να βελτιωθεί. Και θα θέλαμε να δούμε περισσότερη ενθάρρυνση και όχι τόσο έναν τιμωρητικό τόνο. Για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, ε, τρόφιμα και τρίτος κόσμος, το έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Πιο συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική δεν προσφέρει επιδοτήσεις εξαγωγών για τρόφιμα. Κάτι το οποίο ζητούσε ο τρίτος κόσμος για πολύ καιρό. Έπειτα, η ΚΑΠ δεν στρεβλώνει την κατάσταση έπειτα είμαστε μεγαλύτερη εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Έπειτα, οι εταίροι μας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μας το ζητούν και γι' αυτό και ακολουθούμε τώρα μία πολιτική που είναι προσανατολισμένη στην αγορά. Δηλαδή, οι αγρότες παράγουν αυτό το οποίο ζητάνε οι αγορές και όχι που τους ζητούν οι νομοθέτες. Αυτό το ζητούσαν όλοι οι εταίροι μας και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Σε βαθμό που οι τιμές μας τώρα είναι τιμές παγκόσμιας αγοράς όσον αφορά τα αγαθά. Και όχι όπως γινόταν παλιότερα. Δεν γίνεται dumping προϊόντων στην Αφρική. Αυτές είναι ιστορίες του παρελθόντος. Το κείμενο λέει να σταματήσουν κάποιοι μύθοι. Ε, ένας τέτοιος μύθος είναι που λέει ότι εμείς κάνουμε dumping σε τιμές πουλερικών ε, και άλλων προϊόντων. Δεν ισχύει αυτό. Αν δείτε τις εξαγωγές, θα δείτε ότι όλες είναι σε αναπτυγμένες αγορές και υψηλή αξίας προϊόντα. Πολύ λίγα εξάγουμε στην υποσαχάρια ε, Αφρική και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ε, δεν υπάρχει και ζήτηση από αυτές τις χώρες. Υπάρχουν ε, προβλήματα με τα παιδιά, ε, υπάρχουν ε, προβλήματα με προϊόντα πρωτεϊνούχα και γι' αυτό χρειάζονται είτε από την Ευρώπη είτε από άλλες χώρες γιατί δεν υπάρχει προσφορά επιτόπου για τέτοια προϊόντα, γαλακτοκομικά για παράδειγμα και άλλα πρωτεϊνούχα. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στην Αφρική και αλλού οφείλονται σε έλλειψη οργάνωσης, υποδομών. Όλα αυτά είναι πράγματα που εμποδίζουν την ε, εγχώρια παραγωγή αυτές τις χώρες. Και εμείς μέσω της αναπτυξιακής μας πολιτικής, μέσω συνεργασίας, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ζωή μικρών επιχειρηματιών ανά την Εφρική, ώστε να μπουν στην αλυσίδα αξιών στηρίζεται ιδεολογική παραγωγή, ε, προϊόντα υψηλότερη αξίας. Για παράδειγμα, τα φεστίκια κάστους να πηγαίνουν στην Κίνα να ψήνονται πριν έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι βέβαια βιώσιμη πολιτική. Αυτό θέλουμε να αλλάξει. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία κάπως σύντομα για να μπω στο αναφέρει το κείμενό σας. Η γνωμοδότηση επικρίνει το γεγονός ότι στο γαλακτοκομικό τομέα, τομέα για παράδειγμα, εκθέτουμε την ευρωπαϊκή αγορά στην ε, διεθνή αγορά. Δεν ζητούμε συγγνώμηση γι' αυτό. Έπειτα, το κείμενο λέει ότι παρεμβαίνουμε σε θελοντική βάση με την συνδεδεμένη στήριξη. Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε. Θα παρεμβαίνουμε στην αγορά ή δεν θα παρεμβαίνουμε. Από ό,τι φαίνεται λέτε ότι το ένα κάνουμε τι το άλλο κάνουμε, κακώ κάνουμε. Πολύ θα θέλαμε λοιπόν το κείμενό σα να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νέα κοινή γεωργική πολιτική να συνεχίσει την μεταρρύθμιση για ακόμα περισσότερο προσανατολισμό στι αγορέ. Αυτό θα αποφύγει τι τρευλώσει είτε στην Ευρώπη είτε στη διεθνή γεωργία και στι διεθνεί αγορέ. Και ολοκληρώνω με αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Δεν είναι τέλεια η κοινή γεωργική πολιτική, το αναγνωρίζουμε και στην επόμενη μεταρρύθμιση θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται και στις συνθήκες και τους ε, βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Ελπίζουμε και προσδοκούμε όλοι αυτοί να συμπεριληφθούν στον επόμενο εξυγχρονισμό της ΚΑΠ, ώστε αυτοί να καταστεί ακόμα περισσότερο βιώσιμη και ακόμα περισσότερο στραμμένη στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Θα δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε και να θέσετε ίσως ερωτήσεις, αλλά να δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, Μάικλ Κνόπ. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είναι εδώ παρούσα για να υποστηρίξει όσα μόλις εξήγησαν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Γνωρίζετε ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ συνεργαζόμαστε μάλλον πολύ στενά. Συμφωνούμε απολύτως με όσα ακούστηκαν για την ανάλυση που κάνουμε στην ε, αλυσίδα αξίας ε, και ότι στις χώρες που μας ενδιαφέρει περισσότερο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή της εστιάζουμε και ε, συμμετέχουμε από κοινού σε διάφορες τεχνικές ομάδες ε, για διάφορα αγαθά ε, με συναδέλφους από τις χώρες ΑΚΕ για τη ζάχαρη, τις μπαντάνες. Οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας αναφέρθηκαν και στην μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τη διατροφή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα επ' αυτού ε, πράγματι λοιπόν προσπαθούμε μαζί να βεβαιωθούμε ότι θα διασκεδάσουμε τις ανησυχίες των μελών και σίγουρα όλα αυτά είναι εν εξελίξη. Είμαστε απόλυτα αποπισμένοι από κοινού ότι με την ευθυγράμμιση βεβαίως ε, και των εταίρων στις χώρες που θέλετε να υποστηρίξετε, που είναι και το εφαλτήριο σε όλες τις πολιτικές ανάπτυξης, όπως ίσως θα γνωρίζετε. Έχουμε 100 χώρες, τις οποίες υπάρχουν συμφωνίες ανάπτυξιακής βοήθειας. 60 εξ αυτών συμμετέχουν και στους τομείς της γεωργίας. Και με αυτές τις χώρες, όταν ο πολιτικός διάλογος φτάνει μέχρι εκεί που θα ήθελαν όλοι οι εταίροι, σίγουρα μπορεί να επιτευχθεί κάποια πρόοδος ε, με τους εταίρους αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για να ολοκληρώσει ή να θέσει και κάποια ερώτηση, ο λόγος στην συντάκτη. Ε, δεν μου έγιναν ερωτήσεις. Ε, εγώ πρέπει να πω ότι αυτά που ελέγξαν μ' άφησαν εννοεί. τι είναι αυτά. Αυτά που ακούσαμε ε, πραγματικά ε, ελέγχθησαν ε, λόγω αμάθειας. Δεν θα το έλεγα, αλλά αυτή τη φορά προκλήθηκα. Αμάθεια και άγνοια του τι διαδραματίζεται. Ε, τα στρεβλώνετε τα πράγματα και την κατάσταση και θέλω να σας πω αυτά που λέτε είναι του προχθές. Εγώ απευθύνθηκα στον Επίτροπο και του ρώτησα τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις μετακινήσεις. Ε, ε, ο κύριος Χόγαν μου είπε τίποτα, θα αλλάξουμε μια χαρά τα κάνουμε. Και εσείς είπατε σήμερα τα ίδια. Με αυτή την πολιτική ντρέπομαι εγώ ντρέπομαι για αυτά τα οποία είπατε εσείς εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, κάτω του μηδενός, κάτω από οποιοδήποτε ανοιχτό επίπεδο. Μα δεν έχετε καταλάβει ότι οποιαδήποτε μορφή επιδότησης ε, ανάλογα με την έκταση είναι κατ' ουσίαν έμεσα μία χρηματοδότηση των ολίγων. Πραγματικά με αφήνει ενεή η άγνοια σας επί του θέματος. Και αν τελικά απορριφθεί η γνωμοδότησή μου, καλύτερα να απορριφθεί ε, παρά να είναι σε τελική ανάλυση ένα νοθευμένο χαρτί που δεν θα αξίζει ούτε για χαρτί. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ε, προσπαθώ λίγο να δω και πού είμαστε. Πού είμαστε, Ντονατάλα. Υπάρχουν ερωτήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Συγγνώμη γιατί δεν άκουσα. Δεν πρόλαβα φορές ακουστικά. Δεν ξέρω καν τι είπατε. Αλλά δεν φαίνεται και πολύ ικανοποιημένη η συνάδελφος. Θέλετε να απαντήσετε κάτι στην κυρία Νόχελ δεν είμαι δημοκρατικά εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλεύου. δεν μπορώ να έχω το τελευταίο λόγο. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει ε, ενισχύσει εξαγωγών σε καμία χώρα για κανένα προϊόν. Εμείς έχουμε το πράσινο κουτί, βάση του ορισμού του ΠΟΕ. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ε, οι τιμές μας είναι οι παγκόσμιες τιμές της αγοράς. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε και δεν υπάρχει ενίσχυση για αυτές τις τιμές. Ωραία. Μαρία, αν θέλεις να πεις κάτι, όχι. Εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, ούτως ή άλλως ε, ξέρουμε ότι είναι υπάλληλοι οι συνάδελφοι. Μπορούμε να κάνουμε τις συζητήσεις λοιπόν με τους εταίρους μας και τους ε, επιτρόπους. Τελείωσε λοιπόν το σημείο αυτό. Ωραία. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 3η 10 Απριλίου 10 η ώρα και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΔΕΒΕ στις 24 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για το σημείο αυτό. Και τώρα περνάμε στο σημείο 17. Η ώρα των ερωτήσεων. Μία ερώτηση λάβαμε για αυτή τη συνεδρίαση από τον Ιγνάτσιο Κοράου. Θα τη βρείτε στους φακέλους σας. Δεν θα διαβάσουμε την ερώτηση. Μπορείς να μας πεις σε ένα λεπτό περί τίνος πρόκειται και μετά θα απαντήσουν. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν και εγώ είχα χρόνο να το διαβάσω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Είναι αρκετά σύντομη ούτως ή άλλως η η ερωτηση Θα τα καταφέρουμε σε ένα-δύο λεπτά, ξεμπερδεύουμε στην ερώτησή μας εξηγούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγέα και καταναλωτής καφέ και κακάο στον κόσμο. Δύο προϊόντα τα οποία απασχολούν δεκάδες ε, εκατομμύρια ε, γεωργούς και πολλού ανηλίκους. Πληρώνει 60% λιγότερο σε σχέση με το 1983 Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμέ που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κακάο είναι λιγότερο από το μισό των εισαγωγών και δεν μπορεί να ε, εγγυηθεί ε, βιώσιμο εισόδημα. Μην διαβάζετε την ερώτηση σας παρακαλώ. Ναι, αλλά υπάρχουν στοιχεία, άμα δεν τα διαβάζω τα στοιχεία, δεν μπορώ να σας ε, εξηγήσω τι περί τίνος πρόκειται. Είναι στοιχεία, γι' αυτό ακριβώς τα διαβάζω. Θα είμαι σύντομος. Καταγγέλνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη μεταξύ καλλιεργητών καφέ και κακάο που εκμεταλλεύεται την εργασία ε, των ανηλίκων και την απόλυτη φτώχεια. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που δήλωσαν ότι η πιστοποίηση κακάο και καφέ, όπως για παράδειγμα το fair trade κλπ, ε, συνεισφέρουν στις συνθήκες ένδυας και πείνας ε, και κυρίως για τους ανάλικους και τα συστήματα πιστοποίησης λαμβάνουν ε, εκατομμύρια ευρώ ενισχύσει και έτσι οι πολυεθνικέ μπορούν να αγοράσουν κακάο και καφέ σε πολύ χαμηλότερη τιμή από το κόστο παραγωγή και έτσι ε, παραπλανούν και του Ευρωπαίου καταναλωτέ ε, με ψευδεί δηλώσει. Τι μέτρα άμεσα σκοπεύει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει εργασία ανηλίκων στην αλυσίδα κακάο και καφέ που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύσουμε εκατομμύρια ανηλίκου ε, για τι εμπορικέ πρακτικέ που εφαρμόζουν οι πολυεθνικέ ε, και πώ σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί οι καταναλωτέ καφέ και κακάο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συμβάλλουν στη χρηματοδότηση ε, πρακτικών που σχετίζονται με εκμετάλλευση. Δεν μακρηγόρησα και τόσο πολύ. Okay, um, have got the commission to Μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω το όνομά σας δυστυχώς. Η κυρία Ρώσα Α, για τη Γενική Διεθνή Στεύκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Πουλευτά. Εξετάσαμε προσεκτικά το ερώτημα όταν το λάβαμε το Δεκέμβριο και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις ε, μεταξύ των υπηρεσιών μας ε, εκκρεμεί η δημοσίευση και είναι προσεχής. Θα ήθελα να σας διαφάσω όμως ε, τι προτείναμε ε, ως απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εκριζώσει όλες τις μορφές ε, παιδικής εργασίας ε, βάσει και του στόχου του θεματολογίου του 2030 της βιώσιμης ανάπτυξης του αντιστοίχου. Η πολιτική αυτή λοιπόν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για υπεύθυνε αλυσίδε ε, προμηθειών, ε, οι οποίε συμμορφούνται και σε περιβαλλοντικά πρότυπα ε, και λαμβάνουν υπόψη του και θέματα παιδική εργασία σε μη ευρωπαϊκέ χώρε. Διότι η ερώτησή σα δεν διευκρίνει ακριβώ σε ποιε περιοχές ε, διαπιστώνεται παιδική εργασία. Περαιτέρω, εμείς υποστηρίζουμε μέσω και του νομικού πλαισίου με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η γεωργία και φυσικά ε, εργαλεία εμπορίου. Για παράδειγμα, χώρες οι οποίες εντάσσονται στο GSPC, στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, πρέπει να κυρώσουν και να εφαρμόσουν ε, τα θεμελιώδη ε, πρότυπα εργασίας που περιλαμβάνουν και την παιδική εργασία. Τα συστήματα πιστοποίησης στόχο έχουν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των διαφόρων κοινοτήτων, καθορίζοντας κοινωνικών, οικονομικών και ε, περιβαλλοντικών προτύπων, ώστε να γιόμαστε και ότι τα προϊόντα τους πολλούνται σε μια συμφωνημένη ελάχιστη τιμή, που για την περίπτωση του κακάο είναι ε, πάνω από τις τιμές της αγοράς αυτή τη στιγμή. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις ε, για να αυξήσουμε την ε, επιρροή αυτών των προγραμμάτων πιστοποίησης, να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών και των συνθήκων τους διαβίωσης και γίνεται μια μελέτη αυτή τη στιγμή στην ακτή του Ελεφαντοστούν για να δούμε τι γίνεται με τα πιστοποιημένα προγράμματα και τα κλασικά προγράμματα και λογικά θα έχουμε διαθέσιμα τα αποτελέσματα σύντομα και θα ενημερώσουμε για τυχόν μελλοντικέ παρεμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο μέσω ενός εργαστηρίου αύριο κιόλας, 21 Μαρτίου. Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αυτό το εργαστήριο και είστε ευπρόσδεκτοι. Βεβαίως σας καλούμε και υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων από θεσμικά όργανα, από τον ιδιωτικό τομέα, από την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμοί ε, στον τομέα του κακάο. Έχω και κάποιες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εδώ, αν θέλετε, και στο τραπέζι εκεί θα βρείτε αντίγραφα. Και στο εργαστήριο αυτό με χαρά σας ενημερώνω ότι έχουμε προσκαλέσει ως ομιλητή μεταξύ άλλων πέντε ομιλητών και τον κύριο Φορνάντο Μοράλες Τελακρούθ, ο οποίος ε, σας ενημέρωσε ε, για το πρόβλημα. Οι τιμές ε, για τον καφέ και το κακάο ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε διεθνές επίπεδο. Όμως το πρόβλημα του χαμηλού επίπεδου στις παγκόσμιες τιμές ε, καφέ και κακάο θα πρέπει να εξεταστεί κυρίως για τις μεγάλες σύγχρονες εκμεταλλεύσεις. Ένα καλύτερο εισόδημα για του χρήστε, σίγουρα θα βελτιώσει το βιωτικό τους επίπεδο και θα δεν θα υπάρχει εμπλοκή παιδιών σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, υπάρχει και σχετική οδηγία για αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, του 2005, η οποία εξασφαλίζει ότι ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτές ε, για τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύονται προϊόντα κακάο και καφέ. Διότι η οδηγία αυτή μπορεί να απαγορεύσει παραπλανητικές ή ψευδείς ισχυρισμούς στις διαφημίσεις. η εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι ισχυρισμοί κλπ. στις ετικέτες θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς, συγκεκριμένοι και ακριβείς και οι έμποροι θα πρέπει να προσκομίζουν και αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους. Είναι αρμοδιότητα βεβαίως των εθνικών αρχών να αξιολογήσει κατά πόσον κάποιος ισχυρισμός είναι παραπλανητικός είτε ως προς το περιεχόμενο είτε ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στους καταναλωτές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ε, στον τομέα της υφαντουργίας ε, και του Βάμπακα και υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και το ΦΑΟ και θέλουμε να υποστηρίξουμε και μια πρωτοβουλία για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την ειχνηλισιμότητα στις αλυσίδες αξιών. Όταν λοιπόν θα έχουμε τα αποτελέσματα και πιο από τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε ίσως να επαναλάβουμε αντίστοιχη μελέτη και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα του καφέ και του κακάου. Ωραία. Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να ρωτήσετε, Γνάτσιο. Ναι. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη στην οποία αναφερθήκατε και από τη συνάντηση η οποία θα γίνει αύριο, ε, κατά την άποψή μου υπάρχει ένα θέμα ουσίας άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και δύσκολα μπορούμε να βρούμε άμεσες απαντήσεις. Εδώ συζητούμε τον καφέ και το κακάο, αλλά το ίδιο πρόβλημα αφορά και άλλους τομείς. Είναι σαφές ότι η παγκοσμιοποίηση, το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός, ότι μειώνονται οι τιμές για να είναι κάποιος ε, συνέχεια πιο ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυτές τις συνέπειες. Εμείς θα πρέπει να βιαστούμε για να προσπαθήσουμε να προσδώσουμε μια νέα ισορροπία σε αυτό το μηχανισμό τιμών και παγκοσμιοποίηση, διότι είναι σαφές ότι δεν είναι βιώσιμο και κάποιο πληρώνει το τίμημα ε, όταν είναι τόσο χαμηλή η τιμή της αγοράς. Ε, ελπίζω από αυτή τη μελέτη, από αυτή τη συνάντηση αύριο, να υπάρξει συγκεκριμένη δράση στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι για πολλωστή φορά ακούμε πάρα πολύ ωραία λόγια, πάρα πολύ ωραία προγράμματα, αλλά πολύ δύσκολα καταφέρνουμε να δούμε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα μπορέσουν πραγματικά να προφυλάξουν το κόστος της εργασίας, την τιμή της εργασίας και την εκμετάλλευση των παιδιών σε πολλές περιοχές του κόσμου, στις οποίες δραστηριοποιούνται ευρωπαϊκές πολυεθνικές και μέσω αυτών μπορούν να επιτρέψουν σε αυτές τις αγορές με υπερανταγωνιστικές τιμές. Ελπίζουμε να έχουμε πρόοδο και θα παρακολουθούμε και ως Ευρωβουλευτές αιρετή ε, την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θα παρακολουθήσουμε από κοντά την υπόθεση. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή. Στην αρχή τη συνάντηση είπα, χτες δηλαδή, ότι θα έχουμε κάποιου προσκεκλημένου. Θα προσπαθήσουμε 10 λεπτά το πολύ να συνομιλήσουμε με τους ε, προσκεκλημένους μας από την Γουατεμάλα. Έχουμε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Λετήθια Βιλγκουάριο. Η Υπουργό θέλει να μας εξηγήσει ποια είναι η στρατηγική και οι μηχανισμοί συνεργασίας που έχουν να κάνουν με την εθνική πολιτική απασχόλησης στη Γουατεμάλα. Βρήκατε τη διερμηνία, έτσι. Ωραία. Δύο πράγματα θέλω να σας υπενθυμίσω. Το ένα είναι ότι από το δικό μας έργο ελέγχου έχουμε δει ότι τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά, ένα μόνο μικρό τμήμα των κονδυλίων που απευθύνονταν στην Γουατεμάλα έχει εκταμιευθεί. Και θέλουμε να ξέρουμε γιατί. Γιατί είναι κρίμα όταν υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα να μην δαπανούνται τελικά. Θα έπρεπε λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό. Και το δεύτερο είναι να πω ότι τρει υποψήφοι, ε, μία από τους τρει υποψηφίους μάλλον του επικρατέστερους για το βραβείο Ζαχάροφ ήταν από την Γουατεμάλα, ε, γιατί αγωνίστηκε τα, για τα δικαιώματα των ε, αυτοχθόνων πληθυσμών. Βρίσκεται στην Ευρώπη για να προστατευτεί από επιθέσεις, γιατί υπάρχουν απειλές κατά τη ζωή της ε, στη Γουατεμάλα και συνεχίζει το έργο της σε ασφαλέστερες συνθήκες εδώ. Ελπίζω να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στις αρχές της χώρας σας. Εμείς είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύουμε ότι κάποιος που αγωνίζεται για αυτά πρέπει να μπορεί να δρά ελεύθερα. Λοιπόν, λυπάμαι που σας συναντάμε τόσο αργά και για τόσο λίγο, αλλά παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τις 6.30 γιατί θα σταματήσουν οι διερμηνείς. Και εγώ πρέπει να πάω να ψηφίσω σε κάποια άλλη αίθουσα. Οπότε παρακαλώ πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Εκ μέρους της κυβέρνησης της Βατεμάλα, εκ μέρους του κύριου Τζιμοράλες, σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας μέσω του Στέφανου Γκάτο, του πρέσβη σα, για τα στρατηγικά προγράμματα που είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την απασχόληση για όλους εξίσου. Επίσης, ευχαριστούμε και για την βοήθειά σας προς τη Γουατεμάλα όσον αφορά την καταπολέμηση της ατιμορρησίας και της διαφθοράς. Εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθήσατε πολύ, μας στείλατε τα σωστά μηνύματα προκειμένου να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες από πλευράς των αρχών της Βατεμάλας. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω επίσης ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δουλέψει πολύ για να καταπολεμηθούν και οι ανισότητες στη χώρα μου. Οπότε σε σχέση με το τελευταίο που είχε να κάνει με την προστασία μιας γυναίκας ε, αυτόχθονας τη Λολίτα Τσάβες που γνωρίζω, Χαίρομαι για την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αγώνα της όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι κάτι που αναγνωρίζει και η κυβέρνηση της Γουατεμάλα. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι η Δημόσια Εισαγγελία είχε ειδικού πόρους ώστε να έχουμε τώρα μια ειδική μονάδα στη χώρα για την προστασία των αγωνιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η περίπτωση της Λολίτας, των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων. Και για μας ήταν πολύ σημαντικός ο συντονισμός ανάμεσα στο, στην εισαγγελία και στο αρμόδιο Υπουργείο για την Προστασία της Λολίτας. Ο πρόεδρος έδωσε προτεραιότητα και θεώρησε πολύ βασικό ζήτημα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ασφάλεια. Και για το δεύτερο που αναφέρατε, για το δημοσιονομικό ζήτημα και την ε, χρήση των κονδυλίων, ξέρετε ότι οι ανάγκες των, ε, του πληθυσμού είναι μεγάλες. Οπότε η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, βασικές υπηρεσίες υγείας, κάτι πολύ βασικό για την αξιοπρέπεια του πληθυσμού, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, στήριξη της υγείας της ασφάλειας και η καταπολέμηση της ε, κακής διατροφής είναι πράγματα τα οποία έχουμε αναλάβει σαν υποχρέωση και εμείς. Οπότε τα κονδύλια τα οποία δώσατε για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές του πληθυσμού, πράγματι βρισκόμαστε σε περίπλοκη κατάσταση, γιατί η χρήση των κονδυλίων είναι πολύ χαμηλή πράγματι. Και είναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι γίνονται οι κατάλληλες προσπάθειες από την κυβέρνηση της χώρας, προκειμένου μέσω του προϋπολογισμού να υπάρχει μια delivery unit, μια μονάδα αποτελεσμάτων δηλαδή, ώστε να τα καταφέρουμε καλύτερα με τη χρήση των κονδυλίων. Όπως γνωρίζετε, η χώρα έχει σαν κύριε προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την ομοθεσία για τις συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, και είναι δύσκολο να, εκμετα... να τόσο εθνικά κονδύλια όσο και από τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν χρήσης κονδυλίων, εκτέλεσης δηλαδή του προϋπολογισμού, που οδηγεί μερικές φορές στην παράλυση, στην ε, μείωση της χρήσης. Οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι οι, προηγούμενοι, οι προηγούμενες αρχές, κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στη φυλακή. Ο προηγούμενος ε, ε, πρόεδρος και άλλοι βασικοί παράγοντες και οι τωρινοί φοβούνται πάρα πολύ να υπογράψουν την εκτέλεση κονδυλίων εξαιτία αυτού του προβλήματος. Συνεπώς, η πρόταση που υπάρχει από την κυβέρνηση της Βατεμόλα είναι να τροποποιηθεί ο νόμος που διέπει τις συμβάσει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, δίνοντας βέβαια μεγάλη σημασία στη διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες. Σας τα λέω αυτό για να ξέρετε ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε επαρκής χρήση των κονδυλίων. Να ξέρετε ότι το φροντίζουμε, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας. Το Κογκρέσο, η κυβέρνηση της Γουατεμάλα και ελπίζουμε και η κοινωνία των πολιτών να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για να εξευρεθούν λύσεις και να υπάρξει βιωσιμότητα όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας. Για μας είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να μας στηρίζει προκειμένου να προχωρήσουμε και εμείς με τις πολιτικές μας και τη στρατηγική μας που οδηγεί στην ανάπτυξη και την ισότητα στη Γουατεμάλα. Και ολοκληρώνω ευχαριστώντας σας όλους για ένα πρόγραμμα το οποίο θέλησε πάρα πολύ τη Γουατεμάλα. Πρόκειται για το πρόγραμμα όσον αφορά την απασχόληση των νέων. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το 70% του πληθυσμού στη Γουατεμάλα είναι νέοι. Και με το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτήσατε, θέλαμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας, ώστε ο πληθυσμός αυτός των νέων, η νεολαία δηλαδή, που ψάχνει ευκαιρίες ανάπτυξης, να μπορέσει να τις βρει. Η Εθνική Πολιτική Απασχόλησης για αξιοπρέπεια είναι κάτι που προχωράει από τη δική μου την αρμοδιότητα και θέλει να συμπεριλάβει και γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, νέους, ε, μετανάστες, που είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες που απαιτούν και περισσότερη βοήθεια από την πλευρά μας. Εκ μέρους της κυβέρνησης της Γουατεμάλα, λοιπόν, θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να καταπολεμάμε την ατιμορρησία, τη διαφθορά και να συνεχίσουμε τα προγράμματα τα βασικά που απαιτεί και η κοινωνία μας προσωπική ανάπτυξη, κοινοτική ανάπτυξη, κυρίως των αυτόχθονων πληθυσμών, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προκλήσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες και οι δυσκολίες πολύ μεγαλύτερες. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Και σας ευχαριστώ εκ μέρους της κυβέρνησής μου για τη στήριξή σας, για το ότι είσαστε ανοιχτοί απέναντί μας και θέλουμε και εμείς να συντονίσουμε τις προσπαθειές μας μαζί σας και το τελευταίο μήνυμα. Η δέσμευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είναι η ένταξη όλων στην ανάπτυξη με ισότητα για όλο τον πληθυσμό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις επεξηγήσεις που μας δώσατε στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας. Να ξέρετε ότι αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα της χώρας σας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να λυθούν τα προβλήματα της χρηματοδότησης, της ασφάλειας, ε, των ε, αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεπώς, Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σύντομη αυτή η συνάντηση, αλλά ήταν γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος της συνεδρίασή μας. Σημείο 18, διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. 21 Μαρτίου, αύριο, ακρόαση για την επιστηστική βοήθεια. Και επόμενη συνάντηση τον Απρίλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Δερμηνείς, λέει